αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα. Έχουμε μαζί μας εκπροσωπώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Επίτροπο Μοσκοβισή. Κύριε Μοσκοβισή, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Προκειμένου να συνομιλήσω μαζί σας για τις τελευταίες αυτές εξελίξεις όσον αφορά το πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας μετά το χθεσινό Eurogroup. Ένα Eurogroup το οποίο κινήθηκε πολύ θετικά, ήταν ένα από τα καλύτερα που είχαμε για το ζήτημα αυτό το τελευταίο διάστημα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το σύνολο της Ευρωζώνης. Την τελευταία φορά που ήρθα να σας μιλήσω για την Ελλάδα επέμεινα στις εξελίξεις που είχαν λάβει χώρα. Αναφέρθηκα στην ανακεφαλοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών της Ελλάδας. Αναφέρθηκα στη μεταρρύθμιση του φόρου προσθέμενης αξίας. Αναφέρθηκα σε μια στρατηγική προκειμένου να επιληθεί το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και αναφέρθηκα επίσης και σε μια συμφωνία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ταμείο ιδιωτικοποίησεων. Και ήδη τότε είχαμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Και σας είχα πει βέβαια ότι υπήρχαν σημαντικές προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε, ανάμεσα στις οποίες είχαμε με τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που έπρεπε να λάβουν χώρα, προτού ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματο μακροοικονομική προσαρμογή. Ένα πρώτο στάδιο λοιπόν ολοκληρώθηκε την Κυριακή με την έγκριση σημαντικών νομοσχεδίων από την Ελλάδα προκειμένου να μεταρρυθμιστεί το ασφαλιστικό σύστημα, να ενοποιηθεί το ασφαλιστικό σύστημα και προκειμένου να μεταρρυθμιστεί επίσης και το φορολογικό σύστημα της χώρας. Οι δύο αυτές σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ενέκρινε η Ελλάδα θα έχουν μια μόνιμη σημαντική επίπτωση, καθότι αντιστοιχούν περίπου στο 2% του ελληνικού, του ελληνικού ΑΕΠ. Κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα σύστημα πιο βιώσιμο, πιο ισχυρό και μέσω των μεταρρυθμίσεων αυτών όλα τα συνταξιδοτικά ταμεία για όλους τους συνταξιούχους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη χρηματοδότηση. Και βέβαια, παράλληλα μπορούμε να διασώσουμε και τα πιο αδύναμα ταμεία. Και κατά αυτόν τον τρόπο όλοι μπορούν να εισφέρουν ισότιμα όσον αφορά τα έσοδα του κράτους. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν το αποτέλεσμα πολλών συζητήσεων που έγιναν έντονα και κράτησαν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν να κάνουν με την συμβολή της ελληνικής πλευράς σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να χαιρετήσω τους ε, επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όλους δηλαδή αυτούς επικεφαλείς και όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλου, οι οποίοι κατέβαλαν σημαντικότες προσπάθειες συνεχώς, βρίσκονται πάρα πολλοί από αυτούς στην Αθήνα, προκειμένου να ξεπεραστούν κάποια σημαντικά προβλήματα. Οι θεσμοί λοιπόν συνεργάστηκαν θετικά. Οι δύο σημαντικές λοιπόν αυτές μεταρρυθμίσεις αποτελούν τμήμα ενός γενικότερου πακέτου μέτρων που έχει να κάνει με τη Δημιουργεί επίσης ενός ανεξάρτητου μηχανισμού για τα έσοδα, ενός μηχανισμού για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και επίσης προβλέπεται και η θέσπιση ενός νέου Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων και Επενδύσεων και βέβαια όλα αυτά αποτελούν προαπαιτούμενα μέτρα, προαπαιτούμενες δράσεις οι οποίες πρέπει να εγκριθούν. Αυτό το οποίο ζητάμε ουσιαστικά είναι το ότι καταρχάς προφανώς όλα αυτά τα μέτρα θα συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε είναι ακριβώς αυτό. Εδώ και έξι χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε όλες αυτές τις προσαρμογές με απότερο στόχο η ελληνική οικονομία να εξηγιανθεί, τα δημόσια οικονομικά να είναι πιο ισχυρά και να επανέλθει η ανταγωνιστικότητα στη χώρα να έχουμε εκ νέου οικονομική ανάπτυξη και οι επενδυτές να αρχίσουν πάλι να εμπιστεύονται την Ελλάδα. Μια ανοιχτή οικονομία που θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις. Βλέπετε επίσης ότι η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη από το δεύτερο ήμιση του έτους θα παρουσιάσει θετικό πρόσημο. Επίσης θα περάσουμε στο 3% το δημόσιο έλλειμμα το 2017 και Το 2017 θα μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη 2,7% αρκεί βέβαια μεταρρυθμίσεις αυτές να εγκριθούν και ακριβώς για αυτό το λόγο είπαμε ότι ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικό οι μεταρρυθμίσεις αυτές να ολοκληρωθούν και να εγκριθούν. Το μεγάλο κεκτημένο λοιπόν της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup είναι ότι λέμε ναι, επιτέλους οι διαπραγματεύσεις αυτές ολοκληρώνονται, καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, υπολείπονται κάποιες μικρές μόνο λεπτομέρειες και κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να ανακάμψει εκ νέου και θα μπορέσει να οδηγηθεί σε οικονομική ανάπτυξη Ελλάδα. Υπήρχε και ένα δεύτερο τμήμα ζητημάτων που συζητήσαμε και χθε και τις προηγούμενες εβδομάδες, να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία όσον αφορά ένα μηχανισμό δημοσιονομικών μέτρων, έναν έκτακτο μηχανισμό δημοσιονομικών μέτρων. Ο μηχανισμός λοιπόν αυτός που ήδη είχε συζητηθεί στο Άμστερνταμ πριν από μερικές ημέρες θα πρέπει να είναι αξιόπιστο και θα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα. Περί πρόκειται πιο συγκεκριμένα. Θέλουμε να καταφέρουμε να αποκριθούμε σε ένα στόχο που ετέθη από το EMU πέρυσι, να καταφέρουμε να έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 2018. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα τα οποία έχουν εγκριθεί ήδη αρκούν προκειμένου να πετύχουμε το στόχο αυτό πρωτογενούς πλεονάσματος. Παράλληλα όμως δεν συμμερίζονται όλη την άποψη αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν συζητώντας με τα υπόλοιπα μέρη του Eurogroup είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος έκτακτος μηχανισμός προκειμένου να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε όλους τους εταίρους για την αξιοπιστία των δεσμεύσεων της ελληνικής πλευράς. Δηλαδή αν δεν πετυχαίναμε το πρωτογενέ πλεόνασμα, τότε ο αυτόματος αυτός μηχανισμός θα μας διασφάλιζε σε κάθε περίπτωση ότι θα ληφθούν δηλαδή τα επιπλέον αυτά μέτρα προκειμένου να πετύχουμε το πρωτογενές αυτό πλεόνασμα. Καταφέραμε και επ' αυτού να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Επομένως, συμφωνήσαμε και για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, για το πακέτο των μέτρων που έχει εγκριθεί και επίσης συμφωνήσαμε, υπολείπονται μόνο κάποιες λεπτομέρειες και για αυτό τον επιπλέον έκτατο μηχανισμό δημοσιονομικών μέτρων. Επομένως, το μήνυμα το οποίο στέλνουμε σήμερα είναι ξεκάθαρο. Η Ελλάδα με τους εταίρους της κατάφερε να σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο από τον Αύγουστο του 2015 μέχρι σήμερα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον τερματισμό, αν θέλετε. Τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Είναι πολύ σημαντικό τα μέτρα τα οποία πολύ γρήγορα σα παρουσίασα να ψηφιστούν τι επόμενε εβδομάδε. Αυτό αποτελεί προπόθεση προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματο και να εκταμιευτεί και η επόμενη δόση. Προβλέπετε ότι ε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός σταθερότητα θα δώσει ένα σημαντικό ποσό που θα καλύπτει και τις δενειακέ ανάγκες, αλλά επίση και τα ληξιπρόθεσμα ωφέλη του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι θα οδηγηθούμε σε πιο θετικά αποτελέσματα. Και όπω είπε χθε και ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ο επικεφαλή του ESM, είναι πολύ σημαντικό να επιλύσουμε και οποιοδήποτε θέμα ρευστότητα μπορεί να προκύψει. Τέλος, όσον αφορά το τρίτο πακέτο μέτρων, δηλαδή το χρέος. Το ζήτημα αυτό ετέθη από τα κράτη-μέλη και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ως προς αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τη δήλωση που εγκρίθηκε χθε. Ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Ντάισελμπλουμ, είπε ότι θα πρέπει να κινηθούμε σταδιακά. Καταρχά, υπάρχει πρόθεσμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέχρι το 2018 χωρί να αλλάξουμε το πρόγραμμα και χωρί haircut, χωρί να υπάρχει κούρεμα του χρέου. Και στη συνέχεια θα πρέπει να κινηθούμε μεσοπρόθεσμα μετά το 2018 δηλαδή. Να δούμε δηλαδή τότε εάν και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Και τέλος υπάρχει και το μακροπρόθεσμο στάδιο, μετά από κάποιες δεκαετίες δηλαδή, να δούμε ποια άλλα μέτρα θα μπορούσαμε να πάρουμε προκειμένου το χρέος να καταστεί βιώσιμο χωρίς όμως να προβλέπεται απομείωση του χρέους. Το ζήτημα του ελληνικού χρέους είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Αποτελεί κέριο σημείο της συμφωνίας που συνήχθη πέρυσι και χαίρομαι πάρα πολύ που για πρώτη φορά στο Eurogroup έγινε επικοδομητική και ανοιχτή συζήτηση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συμβάλλει από τεχνικής πλευράς σε όλες τις συζητήσεις που θα λάβουν χώρα στο μέλλον. Και όπως συμφωνήθηκε και χθε, οι ελληνικέ αρχές και οι θεσμοί πρόκειται στο μέλλον και τις επόμενες ημέρες να εργαστούν εντατικά προκειμένου να ολοκληρώσουν τη συμφωνία. Είμαι πεπισμένο ότι θα καταφέρουμε στην επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup 24 Μαΐου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Ποια συμφωνία θα είναι αυτή. Καταρχάς έχουμε τα δύο αυτά πρώτα τμήματα τα οποία εξέθεσα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επόμενη εκταμείευση του προγράμματος και έπειτα υπάρχει και το τρίτο τμήμα, το χρέος δηλαδή, ένας οδικός χάρτης για το χρέος. Τα τρία αυτά ζητήματα είναι πολύ σημαντικό από κοινού να αντιμετωπιστούν και από κοινού να έχουμε μια συμφωνία. Χθε με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ είπαμε ότι ε, θα μπορούσαμε να κινηθούμε είτε στον έναν είτε στον άλλο δρόμο, αλλά ήταν σημαντικό να καταφέρουμε από κοινού να καλύψουμε και τα τρία αυτά ζητήματα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τι ελληνικέ αρχέ να ανταποκριθούν στι δεσμεύσει του, προκειμένου να καταφέρουν να έχουν σύντομα την επόμενη δόση. Και μετά τι 24 Μαου θα ξανάρθω εδώ, προκειμένου να σας παρουσιάσω, ελπίζω, μια σφαιρική συμφωνία η οποία θα ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η Ελλάδα και που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επιστρέψει στην οικονομική ανάπτυξη, που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτά τα αγωγικά λόγια είχα να σας πω στην αρχή της συζήτησης αυτής και προφανώς είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε περισσότερο τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες. Μπορώ όμως ήδη από τώρα να σας πω ότι είμαι πεπισμένος, βαθιά πεπισμένος, ότι μετά από τόσες πολλές προσπάθειες και μια κοινή δουλειά που έγινε, κινούμαστε πλέον στη σωστή οδό, στο σωστό δρόμο και πολύ σύντομα θα γυρθούμε σε μια επιτυχή λύση την οποία ελπίζω ότι θα δούμε στην επόμενη συνεδρίαση του ε, Eurogroup ε, η οποία θα αποτελέσει, θεωρώ, ένα ορόσημο όσον αφορά τη θετική εξέλιξη του ε, ελληνικού προγράμματος. Άλλωστε, η ενάτη Μαΐου, όπως ξέρετε, είναι και η γιορτή της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δούμε μια θετική εξέλιξη και στο πρόγραμμα της Ελλάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Ξεκινάμε τη συζήτηση με τις πολιτικές ομάδες. Ο πρώτος που θα λάβει τον λόγο είναι ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Παρακαλώ. Αξιότιμη Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Σήμερα συζητάμε για την Ελλάδα, για την κατάσταση στην Ελλάδα και για το πρόγραμμα και έχουμε τους ανθρώπους στο επίκεντρο. Άνθρωποι που υπέστησαν τα πάνδυνα στην Ελλάδα και για να δούμε ποιες είναι και οι προσδοκίες και των ε, Ελλήνων και σε άλλες ε, χώρες της Ευρώπης ε, οι προσδοκίες που υπάρχουν όταν μιλάμε για αυτή την μεταρρύθμιση και αναθεώρηση. Επιθυμώ να ζουν σε ένα κράτος το οποίο θα είναι λειτουργικό, με τα έσοδα τα οποία θα εισπράττει να είναι αποτελεσματικό που να λειτουργεί καλά το κράτος. Η ανάγκη να μπορέσει να μεταρρυθμιστεί η κρατική μηχανή δεν είναι μόνο θέμα ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό. Και το δικαστικό σκέλος πρέπει να λειτουργεί καλύτερα στην Ευρώπη. Κυρίες και κύριοι, έχουμε την επιθυμία των πολιτών. Η κοινωνική ασφάλεια και ασφάλιση να λειτουργεί. Να μπορεί να έχει αηφορία μακροπρόθεσμα, να είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Και συμβαίνει ότι ο Πρωθυπουργό ε, Τσίπρας ε, στην Ελλάδα τοποθετείται ανοιχτά και λέει δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση από τη μεταρρύθμιση των συντάξεων. Πρέπει να υπάρξει μεταρρύθμιση ώστε με τη δημογραφική εξέλιξη να υπάρξει σταθερότητα. Υπάρχει στην Ευρώπη συνολικά η επιθυμία να μην συνεχίσουμε με τα χρέη. Χώρες που έχουν πολλά βάρη από χρέη είναι δυστυχώς οι χώρες που έχουν και σχηρότερες προοπτικές για το μέλλον. Σταθερή προϋπολογισμοί είναι αναγκαιότητα. Να μην ξεπερνούν τα κράτη τις δυνατότητές τους. Και υπάρχει και η επιθυμία στο τέλος τέλος για την ανάπτυξη. Πρέπει να καταστεί σαφέ όπως είπε ο Επίτροπος Μοσκοβισή το θέμα της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό. Έχουμε το πρόγραμμα Juncker. 80 δις ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί. Και έχουμε και ελληνικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Juncker. Και εκεί τα προγράμματα αυτά από το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να προχωρήσουν. Έχουμε επιθυμίες στο τραπέζι και πολλές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν Αλλαγέ, Θέλω να τονίσω ότι αναγνωρίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει είναι πρόθυμη να προχωρήσει. Κυρίε και κύριοι, αυτά τα οποία περιέγραψα για τι επιθυμίε είναι ακριβώ και οι δικοί μα από το Λαϊκό Κόμμα οι επιθυμίε μα για τη μεταρρύθμιση στην Ευρώπη. Με το ΕΛΚ, με τι κυβερνήσει του ΕΛΚ είχαμε κυβερνήσει που προχώρησαν και έκαναν αυτέ τι αλλαγέ ακριβώ. και στέφθηκαν και με επιτυχία. Η Ιρλανδία το 2015 για παράδειγμα είχε υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξη από την Κίνα. Για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ήταν καλύτερη στι επιδόσει τη στην ανάπτυξη η Ιρλανδία από την Κίνα. Ευχαριστούμε τον Έντα Κένι γι' αυτό. Και επίση να δούμε για την υποστήριξη που δόθηκε σε σχέση με τα προγράμματα. Μία χώρα παρέμεινε ε, ε, ως ε, χώρα που έπρεπε να καλύψει τις διαφορές. Η Ελλάδα δυστυχώς. Πολιτικό εκεί ίσω το πρόβλημα και θα πρέπει να δούμε ότι είχαμε και το θέμα τη ανάπτυξη 7% το 2014 ανάπτυξη και πέρσι με την κυβέρνηση Τσίπρα είχαμε μείον 0,2% ποσοστό ανάπτυξης. Δηλαδή είχαμε μια κατάρρευση, μια απομείωση της οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, η πολιτική του Τσίπρα έβλαψε την Ελλάδα. Το τελευταίο πρόγραμμα του Σαμαρά πριν από ένα χρόνο περίπου αν είχε ολοκληρωθεί θα σήμαινε ότι θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει εξοικονομήσει ένα δίσα ακόμα από τα χρέη της. Θα είχε εξοικονομήσει ένα δις. Τώρα τι κάνουμε. Συζητάμε ότι 5,4 ε, δις πρέπει να εξοικονομηθούν. Είναι μεγάλη, τεράστια διαφορά και γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα χαμένο έτος το περσινό έτος για την Ελλάδα με την κυβέρνηση Τσίπρα που έβλαψε συνολικά την Ελλάδα. Κυρίε και κύριοι, ο Τσίπρας ο ίδιος παραδέχθηκε πρόσφατα ότι με αφέλεια ξεκίνησε το έργο του ως Πρωθυπουργός. Μπορώ να πω αφελή συμπεριφορά στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται, ούτε και στην Ευρώπη επιτρέπεται να είμαστε αφελείς. Θέλω να προσθέσω και να πω ότι πολλές από τις υποσχέσεις που έδωσε προεκλογικά ο Τσίπρας δεν τις στήρισε και αποστασιοποιήθηκε από αυτές. Και τώρα ανεξάρτητα από την Ελλάδα πρέπει να πούμε πανευρωπαϊκά προς τους ψηφοφόρους μην πιστεύετε κύριοι τους λαϊκιστές που λένε ότι μπορούμε να παρεκκλίνουμε, μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τα προγράμματα μεταρρύθμισης. Θα είναι αυτό δαπανηρότατο. Κυρίε και κύριοι, τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Ο συμβιβασμό είναι στο τραπέζι. Όλοι πρέπει αυτό, με, με βάση αυτό να προχωρήσουν και να πετύχουμε πολλά. Θέλω να επισημάνω για την Ελλάδα αυτό το οποίο ανέφερε ο Μητσοτάκη, Κυριάκο Μητσοτάκη, επικεφαλή τη αντιπολίτευση, ότι δηλαδή πρέπει να υπάρξει μια στεναρή ηγεσία ώστε να ξεκινήσει μια σαφή πορεία με ένα, σαφή, με ένα σταθερό προπολογισμό για μια σύγχρονη Ελλάδα και την ανάκαμψη. Οι πολίτε στην Ελλάδα μπορούν να βασίζονται ότι η Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα του υποστηρίξει όταν πρόκειται για την έκφραση αλληλεγγύη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δεχθώ μπλε κάρτε μετά τον πρώτο γύρο δηλώσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριο Τζάνι Πιτέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που ξεκίνησε η πρώτη ελληνική κρίση και βρισκόμαστε εκ νέου εδώ πέρα να συζητάμε για την Ελλάδα. Ο κόσμος έχει αλλάξει όμως από τότε. Σε ένα μήνα, στις 23 Ιουνίου, θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό δημοψήφισμα στον Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τη σημαντικότερη κρίση της μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εμείς όμως εδώ, ακόμα εδώ, Ζούμε ένα remake ενός πολύ άσχημου έργου. Επομένως, αγαπητοί συνάδελφοι, τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πω με απόλυτη σαφήνεια είναι ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά επιμένουμε πάρα πολύ εναντίον πάρα πολλές φορές του ίδιου του ελληνικού λαού. Ο ίδιος ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις του η Eurostat, όπως μας το είπε και ο Επίτροπος Μοσκοβισή, τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι προβλεπόταν. Πολλές μεταρρυθμίσεις ήδη έχουν γίνει. Προφανώς θα πρέπει όμως να διασφαλίσουμε και στο μέλλον ότι όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, όπως η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα ή του δικαστικού τομέα. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι που είπε ο κύριος Βέμπερ. Για μένα το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι η Αθήνα, το πρόβλημα ονομάζεται Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το πρόβλημα είναι αυτές οι ακραίες τάσεις που βλέπουμε πάρα πολλές φορές από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο φαίνεται να θέλει να τιμωρήσει την Ελλάδα και δημιουργούν τώρα την έννοια της προληπτικής λιτότητας. Δηλαδή ότι πρέπει ήδη από τώρα οι Έλληνες να εγκρίνουν μέτρα που όπως είπε και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μέτρα τα οποία θα δολοφονούσαν οποιαδήποτε οικονομία. Στην κατάσταση λοιπόν που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, να δημιουργήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο μια νέα κρίση, θα ήταν πραγματικά ανεύθυνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μασκοβισή και γενικότερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χθεσινή του εργασία στο Eurogroup, γιατί αυτή τη στιγμή πληρούνται όλε οι προποθέσει προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματο και να ξεκινήσει επιτέλου και το κεφάλαιο τη ελάφρυνση του χρέου. Δεν λέω απομείωση, λέω ελάφρυνση του χρέου για την οποία δεσμευθήκαμε πριν από ένα χρόνο. Γι' αυτό μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Εμεί εξ αρχή ω Ευρωπαίοι Σοσιαλιστέ ήμασταν πεπισμένοι ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια συμφωνία ανάμεσα σε όλε τι πλευρέ μία ισότιμη συμφωνία που θα έθετε κάποιες ευφυείς μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να κάνει η Αθήνα και από την άλλη όμως θα πρόσφερε στην Αθήνα και ελάφρυνση του χρέους. Αυτή τη στιγμή, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση, δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και πρέπει να πω εδώ πέρα ξεκάθαρα το εξή. Αν το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έρθει να σαμποτάρει για μία ακόμα φορά τη συμφωνία αυτή, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση σύσσωμη θα πρέπει να έχει το κουράγιο και το θάρρος να συνεχίσει μόνη της. Thank you. Κύριος Μαριάς έχει το για δύο λεπτά. Κύριε Μοσκοβισή και κύριε Βέμπερ, πέρασαν έξι χρόνια από τότε που η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια. Έξι πέτρινα χρόνια στα οποία το ΑΕΠ της Ελλάδας μειώθηκε κατά 25%. Το 40% του ελληνικού πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας οι μισθοί και οι συντάξει μειώθηκαν η ανεργία ξεπέρασε τα 1,5 πέντε εκατομμύριο άτομα χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις έκλεισαν η φορολεηλασία της περιουσίας των ελλήνων χτύπησε ταβάνι και το χρέος από 125% του αεπ που ήταν το 2010 φτάνει το 200% του αεπ το 2016. Κι όμως η Τρόικα και ιδίω το Δουνουτού συνεχίζει το business as usual και επέβαλε εν ώψη της ολοκλήρωσης της πρώτης αξιολόγησης επιπλέον μέτρα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ψήφισε η νέο μνημονιακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία σύριζα ανέλ. επίσης επιβάλλει η τρόικα συμπληρωματικά μέτρα κάβα 3,6 δισευρώ, ευρώ συν δημοσιονομικό κόφτη. Έτσι το χθεσινό Eurogroup, κύριε Μοσχοβησή, συνέχισε τη γνωστή αποτυχημένη μνημονιακή πολιτική που επιρρέτησε και η κυβέρνηση Σαμαρά, κύριε Βέμπερ, της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής της περκελική λιτότητας της φορολεηλασίας της μεσαίας τάξης του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και των κόκκινων δανείων. αποτελεί λοιπόν η χθεσινή απόφαση του eurogroup ένα νέο κοινωνικό αρμαγεδόνα ένα μνημείο κινησμού της τρόικας και των δανειστών απέναντι στο φτωχοποιημένο ελληνικό λαό. όσο για τη δίθεν ρύθμιση του χρέους έχουμε επανάληψη του ίδιου έργου άρνηση άμεσης επιστροφής εδώ και τώρα των κερδών της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα που μόνο για το διάστημα 14-16 φτάνει στο 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούσαν να πάνε για την ανάπτυξη. Ξανά λοιπόν υποσχέσεις αβέβαιες, αόριστες για δίθεν μελλοντική διευθέτηση του ελληνικού χρέου, όταν, εάν και εφόσον ενό χρέου που έχει αποδειχθεί κύριε Βέμπερ ότι είναι επονίδιστο αφού από τα 220 δισεκατομμύρια ευρώ είναι odious debt, είναι στο χρέο. Από αυτά τα 220 που δόθηκαν ω δάνεια στην Ελλάδα τα μνημονιακά χρόνια μόνο 9 δισεκατομμύρια ευρώ μπήκαν στα ταμεία και τα υπόλοιπα 214 δισεκατομμύρια ευρώ επέστρεψαν στις τσέπε των δανειστών διασώζοντας τις γερμανικές και άλλε τράπεζε. Φτάνει πια κύριε Μοσκοβισή και κύριε Βέμπερ ο ελληνικός λαός δεν αντέχεται πια τη φτώχεια και δεν ανέχεται την εκμετάλλευση και την ταπείνωση και σύντομα θα πετάξει την τρόικα έξω από την πατρίδα μας για να ξαναπάρει πίσω την ελλάδα. ευχαριστώ. Thank you. Next speaker is Madame Goulard. Η κυρία Γκουλάρ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω τα όσα μα είπατε ότι δηλαδή ήταν επικοδομητικές πλέον οι συζητήσεις στο Eurogroup, ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πιο θετικά, πιο ευίωνα Παρ' όλα αυτά υπάρχει κάτι που με ενοχλεί, γιατί έχω την εντύπωση ότι οι σημερινέ μα συζητήσει είναι συζητήσει ανθρώπων που έχουν γνώση εκ των έσω και βλέπουν τα πράγματα εκ των έσω, έχοντα κάποια τεχνική γνώση των πραγμάτων. Του υπόλοιπου όμω Ευρωπαίου, οι Έλληνε πολίτε, εδώ και έξι χρόνια, το είπαν και οι προαλήσαντε, διανύουμε μία κρίση και κάνουμε συνόδου για την Ελλάδα. Γιατί 9-10 ε, Μαΐου του 2010 ξεκίνησε όλη η ιστορία και εδώ και έξι χρόνια έχουμε και την έκθεση του Μάριου Μόντι για την ενιαία αγορά. Και τι βλέπουμε. Δεν υπάρχουν απαραίτητε επενδύσει, δεν υπάρχει απαραίτητη οικονομική ανάπτυξη. Προσπαθεί το σχέδιο Juncker να επιλύσει τα πράγματα, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε όχι μόνο μια Ευρωζώνη, αλλά μια Ευρωπαϊκή Ένωση 28 κρατών μελών, η οποία δεν πηγαίνει καλά, δεν σημειώνει πρόοδο. Σε όλε αυτέ τι συζητήσει λοιπόν που κάνουμε, δίνουμε την εντύπωση ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ αργά και ότι δεν καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Και όσον αφορά επίσης και την νομιμοποίηση των θεσμών που λαμβάνουν όλες αυτές τις αποφάσεις. Και εκεί δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο. Καταλαβαίνω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά καταλαβαίνω ότι πολλές φορές αναγκάζεται να κάνουμε πράγματα εκτάκτως στην τελευταία στιγμή, αλλά από την άλλη δεν καταφέρνουμε τελικά να δούμε τις θετικές επιπτώσεις ούτε από την έκθεση των πέντε προέδρων, ούτε από το προσχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οικονομική Ανάπτυξη. Όλα αυτά μας δίνουν την εντύπωση τελικά έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία δεν καταφέρνουμε τελικά να ελέγξουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μα και το Brexit, το οποίο θα επηρεάσει τα πράγματα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Και αυτό το οποίο με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν μετά το 2018 και μετά. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, είναι προ το συμφέρον τη Ελλάδα ή το κάνουμε μόνο και μόνο επειδή έχουμε εκλογέ στη Γαλλία και στη Γερμανία. Ο κύριο Παδημούλη, έχει το λόγο για δύο λεπτά. Πρόεδρε, κύριε Βέμπερ, στα πέντε λεφτά τη ομιλία σα επιτεθήκατε πέντε φορές στον έλληνα πρωθυπουργό τον κύριο τσίπρα για να βοηθήσετε τον πολιτικό σας φίλο τον κύριο μητσοτάκη αλλά δυστυχώς η αλήθεια δεν σας βοηθά γιατί οι φίλοι σας της νέας δημοκρατίας άφησαν το 2009 την Ελλάδα με δημόσιο έλλειμμα 15,5% με δημόσιο χρέος 125% του αεπ και στο τέλος του 2014 μαζί με το πασόκ είχαν φτάσει το δημόσιο χρέος στο 180% του αεπ. Μπορεί να βλέπετε κύριε Βέμπερ τον κύριο Τσίπρα ίσως και στον ύπνο σας. Σας βεβαιώνω όμως ότι όπως δεν μπορέσατε να βοηθήσετε τον κύριο Σαμαρά, δεν μπορείτε να βοηθήσετε και τον κύριο Μητσοτάκη. Θα βλέπετε τον κύριο Τσίπρα για πολλά χρόνια ως Πρωθυπουργό, γιατί αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Χτες ήταν μια καλή στιγμή και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη στο eurogroup μετά από έξι χρόνια άγριας σκληρής μονόπλευρης λιτότητας τεράστια ύφεση, τριπλασιασμού της ανεργίας μεγάλης φτώχειας είχαμε επιτέλους κάποιες θετικές ειδήσει που μπορούν να βοηθήσουν την ελλάδα και τον ελληνικό λαό να εξασφαλίσει επιτέλους μεγαλύτερη σταθερότητα πολιτική και οικονομική ταχύτερη επιστροφή στην ανάπτυξη με βάση και τις αισιόδοξες προβλέψεις που έκανε η κομισιόν και ο κύριος Μοσχοβησί και εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ευρωπαίο φορολογούμενο. αλλά είναι μια απόφαση που βοηθά και την ευρώπη να αποφύγει μια αχρίαστη νέα κρίση και αποσταθεροποίηση στον ωκεανατολικό της άκρο όπως προσπάθησε με τα εκβιαστικά παράλογα ανεύθυνα πράγματα που ζητούσε το διεθνές νομισματικό ταμείο χθες το eurogroup απέρριψε τις υπερβολικές και παράλογες απαιτήσεις για νέα πρόσθετα ηφαισιακά μέτρα λιτότητας που ζητούσε το διεθνές νομισματικό ταμείο και χθες το eurogroup χάραξε ένα σαφή οδικό χάρτη για την ουσιαστική ελάφρυνση του δημόσιου χρέους ακυρώνοντας τα σχέδια όσων ήθελαν την αθέτηση αυτής της δέσμευσης. μπροστά μας έχουμε δύο προκλήσεις η ελλάδα θα τιμήσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει για να επιστρέψει το ταχύτερο στην ανάπτυξη κάνοντας όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. αλλά και η ευρώπη η ενωμένη ευρώπη οφείλει να τιμήσει την δέσμευσή της για ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους και να την κάνει συγκεκριμένη και ουσιαστική. σας ευχαριστώ. Κύριος Λάμπερτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο, Γιάν, ο Ζαν Κλοντ μας είχε πει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη είναι εξίσου σημαντική με την δημόσια εξυγίανση και με τους οικονομικούς δείκτες. Από τότε που ξεκίνησε η κρίση και μετά από τα τρία μνημόνια στην Ελλάδα βλέπουμε ότι αυξήθηκε πάρα πολύ ο αριθμός των ε, Ελλήνων οι οποίοι πλήττονται από την κρίση είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι στην αρχή της κρίσης. Πολλοί λένε ότι πρέπει να πληρώσει για τα παρελθόντα λάθη της η Ελλάδα. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, ο χρηματοπιστωτικός τομέας για παράδειγμα, οι εφοπλιστές ή ε, ο τομέας των αμυντικών εξοπλισμών που αποφελήθηκε από την οικονομική αυτή κρίση στην Ελλάδα και δεν καταβάλουν αυτή το τίμημα. Βλέπετε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι ότι εγώ δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του χθεσινού Eurogroup μας δίνει τη δυνατότητα ενδεχομένως να μιλήσουμε για έναν τρόπο ελάφρυνσης του χρέους. Ποιο είναι όμως το τίμημα για τη συζήτηση αυτή. Το τίμημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Τόσο μεγάλο που θεωρώ ότι οι πραγματικές πιθανότητες μείωσης του χρέους, ελάφρυνσης του χρέους, ε, είναι πολύ μικρές. Νομίζω ότι ε, θα έπρεπε ήδη από το 2010 οι πιστωτέ να είχαν αναλάβει τι ευθύνε του, ενώ τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε εν έτη 2016 είναι να τίθενται περισσότερε προποθέσει, να πρέπει δηλαδή να δεχθεί ακόμα περισσότερη λιτότητα η Ελλάδα, προκειμένου να γίνει μια κάποια ελάφρυνση του χρέου. Μια λιτότητα η οποία τονίζεται όλο και περισσότερο ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει πλέον ότι η λιτότητα είναι αντιπαραγωγική. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που ζητά ελάφρυνση από την άλλη του χρέους. Επομένως, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αυτοί οι οποίοι θέλουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην όλη διαπραγμάτευση δεν ακολουθούν από την άλλη τις συστάσεις του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου που ζητά πλέον λιγότερη λιτότητα και μεγαλύτερη ελάφρυνση του χρέους. Προφανώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει κάνει πολλά λάθη και βέβαια αυτά τα λάθη δεν έχουν αναγνωριστεί τη στιγμή που έχουν απέναντί τους βέβαια και μια ελληνική κυβέρνηση που δεν ανήκει στο ίδιο πολιτικό φάσμα με αυτό το οποίο διέπει εν γέννη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. και και το ζήτημα των επενδύσεων που μειώθηκαν κατά 70% στην Ελλάδα από την αρχή της κρίσης. Και όλοι γνωρίζουμε ότι οι επενδυτικές ικανότητες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μηδενικές. Και το μόνο που τους λέμε, λέμε αυτή τη στιγμή προς τους Έλληνες είναι ότι θα σας δώσουμε κάποια ψίχουλα από το επενδυτικό σχέδιο του Juncker. Υπάρχει και επίσης ε, το ζήτημα της δημιουργίας ενός στεναρούς δημοσιονομικού συστήματος. Ξέρω προς αυτό δεν καταβλήθηκαν απαραίτητες προσπάθειες προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να συγκεντρωθούν οι απαραίτητοι φόροι, αλλά νομίζω ότι και οι χώρες της Ευρωζώνης που θα μπορούσαν από τεχνικής πλευράς να είχαν βοηθήσει, τελικά δεν το κάνανε, καθότι πιέσανε για πολύ περισσότερες απολύσεις, επομένως δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό προκειμένου να το στείλουν και στην Ελλάδα. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε μια Ελλάδα η οποία υποφέρει πάρα πολύ, η οποία έχει εγκαταληφθεί απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις, την πρόκληση συγκεκριμένα την προσφυγική και είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ελλάδα να μπορέσει να ανοικοδομηθεί. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσφέρει περισσότερα ανταλλάγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ο κύριος Βούλφ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Το 2001 είπε εγκαινιάζοντας την υιοθέτηση του ευρώ ότι επιτέλους ο Πρωθυπουργό της Ελλάδας θα έχουμε ανάπτυξη, θα έχουμε σταθερότητα, θα έχουμε τη δυνατότητα ευημερία. Ας συγκρίνουμε αυτή τη δήλωση με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. 25% αναργία, 52% η αναργία των νέων. Σκεφτείτε πόσοι νέοι Έλληνες έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους για να βρουν δουλειά στο εξωτερικό. 6.000 αυτοκτονίες. 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε μέτρα λιτότητας. Και θα πρέπει να βρουν τους επόμενους μήνες οι Έλληνες άλλα 5 δισεκατομμύρια να πληρώσουν στους πραγματικούς ε, ε, ε, ελέγχονται στη χώρα τους την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν και το Διεθνές Νομισκό Μαθηματικό Ταμείο. Βοήθησε λοιπόν αυτή η πολιτική. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ο λαός της Ελλάδας αντιτιθέτων ε, στην λιτότητα της δηλώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ε, θυμάμαι ε, τον εναγκαλισμό του Έλληνα Πρωθυπουργού από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θυμάμαι να προσπαθεί να, να ε, υπερασπιστεί το δημοψήφισμα του ελληνικού λαού και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απογοήτευσε τους Έλληνες πολίτες με την πολιτική της. Και σήμερα ακούμε από το ΕΛΚ και από τους σοσιαλιστές να μιλούν για αλληλεγγύη. Βεβαίως, εσείς που ζείτε στην πολυτέλεια μπορείτε να ομιλείτε για ελληνική, αλλά προσπαθήστε να το πείτε σε αυτό στις οικογένειες των 6.000 ανθρώπων που αυτοκτόνησαν. Η κατάσταση στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται. Βλέπουμε ότι η οικονομία έχει συρρυκνωθεί κατά 27% τα τελευταία πέντε χρόνια. Όπως είπε και ο κύριος Πιτέλα, θα έχουμε το δημοψήφισμα στην Μεγάλη Βρετανία για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα μα επιτρέψει να ζούμε καλύτερα, γιατί πλέον δεν θα μα υποβάλουν οι Βρυξέλλε τι αποφάσει του ούτε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ούτε το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Εάν ακούσουμε τις απειλές που εκτοξεύονται ε, ε, στους ε, Έλληνες τους λένε ότι θα φύγουν οι επιχειρήσεις, ότι θα ε, ε, δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερη ανεργία. Εγώ σας λέω ότι εάν η Ελλάδα επιλέξει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως σκοπεύει να το κάνει η Βρετανία στις 23 Ιουνίου, η ζωή των Ελλήνων θα γίνει πολύ καλύτερη. Ο κύριος Ντεγκράφ, επόμενος 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, η Ελλάδα χρεοκόπησε η χώρα είναι ένας ασθενής που κάθε έξι μήνες ε, πρέπει να παίρνει νέο αίμα. Έχει κοστίσει δισεκατομμύρια διάσωση. Τι έγινε με αυτά τα χρήματα. Δέκα δισεκατομμύρια περίπου εντωμεταξύ κατέληξαν στον προϋπολογισμό. 140 δις χρησιμοποιήθηκαν όσον αφορά γαλλικές και γερμανικές τράπεζες που έπρεπε να διασωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ματώνουν, να υφίστανται αφέμαξη λόγω των σφαλμάτων της ευρωπαϊκής ελίτ. Πρόκειται για δισεκατομμύρια τα οποία δεν θα επιστραφούν ποτέ. Πρόκειται για χρήματα τα οποία στην Ολλανδία ε, προσφέρθηκαν και τι συμβαίνει τώρα με όλα αυτά και τι συμβαίνει για τους ε, ηλικιωμένους, ε, για την ασφάλιση, για την, τις συντάξεις, για την ενίσχυση των συνόρων, για μεγαλύτερη ασφάλεια. Και από πλευράς Πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια των εκλογών αναφέρθηκε από μας ε, την, ε, τους Ολλανδούς ούτε δεκάρα πια στην Ελλάδα. Τι μεγάλο ψέμα ήταν αυτό. Ήταν μια πολιτική κατάρρευση αυτή που ακολουθήθηκε με τέτοιου είδους αρχές ε, για να ε, να ε, καλυφθεί, να κρυφθεί ότι είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα και ήταν ασθεν, ένας ασθενής που με ε, τεχνητούς τρόπους τον διατηρούσαμε ζωή. Να μην συνεχίσουμε να περικόπτουμε συντάξεις εις βάρος των πολιτών. Πρέπει η Ελλάδα να μπορέσει να ξαναγυρίσει σε πορεία ανάπτυξης. Φτάνει πια. Στη συνέχεια παρακαλώ θα λάβει τον λόγο ο κυρίος Παπαδάκης. Ένα λεπτό. που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κατεδαφίζει τα ασφαλιστικά δικαιώματα του λαού ενώ γενικεύεται ταυτόχρονα και η άγρια φοροαφέμαξή του. έγκριση από τη βουλή έχετε νομιμοποίηση του λαού για όλα αυτά όμως δεν πήρατε ποτέ. παρά τους ανταγωνισμούς σα, συμφωνείτε όλοι σας ευρωπαϊκή ένωση διεθνές νομισματικό ταμείο και κυβέρνηση ότι κριτήριο για την αξιολόγηση είναι η πάνθινη εργασία και τα προκλητικά προνόμια στο μεγάλο κεφάλαιο αυτή είναι η στρατηγική των μονοπωλίων που υπηρετείται με μόνιμο θύμα το λαό τόσο στην κρίση όσο στην όποια ανάκαμψη έρθει. οι μόνιμοι μηχανισμοί διαδοχικών αντιλαϊκών μέτρων οι αυτόματοι κόφτες μισθών συντάξεων δικαιωμάτων είναι τα μνημόνια διαρκείας της ευρωπαϊκής ένωσης όχι μόνο στην ελλάδα αλλά και σε όλα τα κράτη μέλη της. σε αυτά μπορεί να μπει τέλος εάν μπει στο στόχαστρο η ίδια η καπιταλιστική οικονομία που έχει κριτήριο το κέρδος. ένας αποφασισμένος λαός μπορεί να την ανατρέψει και να γίνει ο ίδιος ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει. Thank ευχαριστούμε. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, μισή λεπτό παρακαλώ τελικά ο winston τσόρτσιλ είχε δίκιο όταν έλεγε αν θες να απαλλαγείς μια για πάντα από την αριστερά τα πρόσθετα και το λαϊκισμό πρέπει να τους αφήσεις να κυβερνήσουν τρεις τέσσερις μήνες. στην περίπτωση της ελλάδος η ουτοπία και οι αυταπάτες όπως παραδέχθηκε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη βουλή στήγησαν στον ελληνικό λαό κάτι παραπάνω. πράγματι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προσδιορίσαν τους στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής για μεν την κυβέρνηση σαμαρά το δεκέμβριο του 2014 στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ για δε την κυβέρνηση τσίπρα τώρα στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ και να προσθέσουμε και 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρα προληπτικής λιτότητας. για τη λύση του ελληνικού προβλήματος η κυβέρνηση τσίπρα επέλεξε τον εύκολο δρόμο το δρόμο της αύξησης της φορολογίας. η υπέρμετρη όμως αύξηση της φορολογίας οδηγεί σε μείωση σε μηδενισμό των δημοσίων εσόδων. το πρόγραμμα κινδυνεύει να μην βγει και τον οκτώβριο να χρειαζόμαστε νέα μέτρα. για το χρέος χρειάζεται ρύθμιση χρειάζεται ελάφρυνση. η ευρώπη έδειξε αλληλεγγύη. μειώθηκε το 2012 το χρέος κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ η εξυπηρέτησή του χρειάζεται 4 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από 16 που χρειαζόταν στο παρελθόν. η κυβέρνηση τσίπρα δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το χρέο ε, ω το τελευταίο φύλλο οική μια αποτυχημένη διαπραγματεύση. η ελλάδα χρειάζεται γιγαντιές δημόσιε και ιδιωτικέ επενδύσει, χρειάζεται να απελευθερώσει όλε τι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου χρειάζεται να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξη για να περάσει αυτή τη μεγάλη και παρατεταμένη κρίση με το μικρότερο δυνατό κόστο. ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Ο κύριος Γουαρτιέρη τώρα, δύο λεπτά παρακαλώ. you, Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς πιστεύω ότι το ελληνικό μνημόνιο του προηγουμένου θέρους είναι πολύ φιλόδοξο στην προσπάθειά του να βρει μια ισοσταθμισμένη προσέγγιση μεταξύ σταθερότητας, ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Θέτει όμως και πολύ μεγάλες απαιτήσει, διότι είναι πολύ ευρύ στο φάσμα του και είναι ιδιαίτερα απαιτητικό. Ταυτόχρονα όμως νομίζω είναι πολύ δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι αυτή η ελληνική κυβέρνηση κάνει τη δουλειά της και έχει σοβαρά δεσμευθεί να ακολουθήσει μεταρρυθμίσεις και να υλοποιήσει τα συμπεφωνημένα. Για αυτούς τους λόγους είναι θετικό ότι επιτέλους καταλήξαμε σε μια συμφωνία για τη δέσμη μέτρων, για τα δημοσιονομικά μέτρα και τα μέτρα στήριξης που είναι αναγκαία για να προχωρήσει το πρόγραμμα και να ολοκληρωθεί. Είναι επίσης θετικό αποτέλεσμα ότι ο μηχανισμός θα βασίζεται στις ελληνικές προτάσεις και δεν θα επιβάλλει στους Έλληνες πολίτες επιπρόσθετα προληπτικά μέτρα λιτότητας που θα ήταν πραγματικά αποσταθεροποιητές. Γνωρίζω ότι το θεσμικό όργανο που ήταν υπέρ αυτής της επιλογής κατέληξε σε προγνώσεις για την οικονομική εξέλιξη που ήταν απόλυτα λανθασμένες αυτές οι προγνώσεις και ελπίζουμε ότι στο τέλος τέλος θα μπορέσει η προοπτική ανάκαμψη να υλοποιηθεί. Καλωσορίζουμε τη συζήτηση για πρόσθετη ανακούφιση χρέους. Και τώρα υπάρχει ένας μύτο της Αριάννης, κατευθυντήριες γραμμές για να ταυτοποιηθούν συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την ε, επέκταση, ε, ώστε αυτή η προσέγγιση, και αυτό είναι ένα άλλο θετικό στοιχείο, να μην αποκλεί περαιτέρω μέτρα μακροπρόθεσμα. Έτσι λοιπόν η 9η Μαΐου πράγματι ήταν μια καλή θετική ημερομηνία για την Ευρώπη. Θετική ημέρα. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή και κυρίω τον Επίτροπο Μοσκοβισή για τον κέριο ρόλο που επετέλεσε και είχε. Τώρα πρέπει να οδηγηθούμε στην 24η Μαΐου ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να ξαναγυρίσει στη διαδρομή ανάπτυξης και σταθερότητας και να αποσταλεί ένα σαφές μήνυμα ότι η Ευρώπη είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια τόσο περίπλοκη και δυσχερή κρίση και μπορεί να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ανάπτυξη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο παρακαλώ ο κύριος Λούκ. Κυρίες και κύριοι, είναι εκπληκτικό να ακούει κανείς εδώ λόγους ε, που στρεβλώνουν τα γεγονότα και τα στοιχεία. Θέλω να υπενθυμίσω ότι πριν από έξι χρόνια ακριβώς ε, με τη μέρα αυτή έξι χρόνια που ε, διεράγησαν οι συνθήκες και άνοιξε αυτή η ε, δυνατότητα προστασίας για την Ελλάδα. Αναφέρθηκε ότι επί τρία χρόνια θα έπαιρνε χρόνια η Ελλάδα, 2013 θα τερματιζόταν αυτή η διαδικασία και θα στεκόταν η Ελλάδα στα πόδια της. Σήμερα έξι χρόνια πέρασαν και δεν στέκεται στα πόδια, τα της η Ελλάδα. Κάνουμε λόγο για το 2016, 17, 18, δεκαετίες ολόκληρες ε, που θα επιβαρύνει τη Ελλάδα με χρέη. Έχει αποτύχει η πολιτική αυτή κυρίες και κύριοι. Και τώρα από πλευράς Επιτροπής όταν γίνεται η επισήμανση ότι βελτιώνονται τα πράγματα, αυτά τα ακούμε επί χρόνια τώρα. Κάθε χρόνια οι προγνώσεις της, επιτροπή Επιτροπής ε, πέφτουν έξω επί, επί διάφορες ποσοστίες μονάδες. Και αναφέρεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει φταίει και όποιος το κάνει αυτό στρεβλώνει την πραγματικότητα. Η Ελλάδα δεν ε, μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική λιτότητα ενώ πριν από τρία χρόνια έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδρομή. Απέτυχε η Ελλάδα, χρεοκόπησε, πρέπει να αποπεμφθεί από τη ζώνη ευρώ ώστε να μπορέσει να γίνει καλύτερη η κατάστασή τη. Ευχαριστώ. Κύριε Λούκε, έχετε μία μπλε κάρτα, μπορείτε να δεχτείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε για την δυνατότητα που μου δίνετε για τρίτη φορά την ευκαιρία να διατυπώσω μια ερώτηση. Αγαπητέ κύριε Λούκε, παρακολούθησα, άκουσα την τοποθέτησή σας και ομοιάζει με τις τοποθετήσεις ε, κάποιων άλλων προλαλισσάντων από, την, από το ΕΛΚΑ. Πώς κατανοείτε την αλληλεγγύη εσείς όμως. Η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις συνθήκες αναφέρεται σαφέστατα ποια είναι και τι είναι η αλληλεγγύη. Εσείς πώς εννοείτε το θέμα της αλληλεγγύης όταν πρέπει να βοηθηθεί ένα κράτος που αντιμετωπίζει προβλήματα. Παρακαλώ απαντήστε. Ο κύριος Λούκε. Κυρία συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας ότι πρέπει να εκφράσουμε αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εκείνους που είναι φτωχοί, που δεν έχουν επαρκείς υποδομές, ε, όπου οι, κοινωνικές, ε, ε, οι κοινωνικοί θεσμοί δεν μπορούν να υποστηριχθούν όπως πρέπει. Όμως δεν πιστεύω κυρία μου ότι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με εκείνους που έριξαν έξω την οικονομία. Δεν πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη με εκείνους που είναι υπερχρεωμένοι. Δεν πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη με εκείνους που τα συμπεφωνημένα μέτρα δεν τα τηρούν από πλευράς προγραμμάτων και εδώ και χρόνια δεν τα εφαρμόζουν πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά οι όροι και οι προϋποθέσεις ε, για να τηρούνται αυτά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε λέγει η Πρόεδρος. <clears throat> Στην ε, συνέχεια παρακαλώ ατουή, δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την Ελλάδα εδώ και έξι χρόνια μας δίνουν ένα θέμα το οποίο είναι τρομακτικό βλέπουμε να επικρατεί ο χρηματοπιστωτικό τομέα και βλέπουμε ότι είναι αδύνατο να ληφθεί μια κάποια απόφαση. Η Ελλάδα έφτασε στο χείλος του γκρεμού και αυτό αποτελεί και δική της βέβαια ευθύνη, διότι ε, παραποίησε δημόσια οικονομικά, αλλά είναι ευθύνη και των ίδιων των πιστωτών. Γιατί ήδη από το 2009 οι πιστωτές της Ελλάδας θα έπρεπε να είχαν συνειδητοποιήσει ότι θα έπρεπε να είχαν μειώσει το χρέος της Ελλάδας, προκειμένου αυτό να γίνει βιώσιμο και προκειμένου οι εθνικές αρχές να μπορέσουν δημοκρατικά να βρουν τις απαραίτητες απαντήσεις, προκειμένου να καταφέρουν να κερδίσουν την ε, εμπιστοσύνη των ε, δανειστών. Ανταυτού είδαμε ότι δημιουργήθηκαν πολύπλοκα συστήματα τα οποία δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη. Πώς μπορούμε να αφήσουμε μια χώρα που έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο είναι το διπλάσιο του ΑΕΠ της αυτή τη στιγμή. Πραγματικά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης δεν τηρείται και αυτό το οποίο βλέπουμε στην πράξη είναι ότι δίνουμε όλο και περισσότερα δάνεια στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να καλύψει τα ληξιπρόθεσμα δάνειά τη. Και κατά αυτόν τον τρόπο διονύζουμε μια κατάσταση που μόνο δραματική κατάληξη θα μπορούσε να έχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε συγκεκριμένε πολιτικέ και ραλιστικέ πλέον αποφάσει. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η χτεσινή απόφαση του eurogroup αποτελεί μνημείο οικονομικής υποτέλειας και επιβολής οικονομικής ισχύω σε βάρος της ελλάδος. χθες εσείς οι υπουργοί της ευρωζώνης υποσχεθήκατε για άλλη μια φορά στην νεομνημονιακή κυβέρνηση μελλοντική διευθέτηση ενός χρέους που δεν διευθετείται και έτσι πετύχατε νέα αντιλαϊκά μέτρα. χτες κύριε επίτροπε και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ο έλληνας υπουργός οικονομικών παρέδωσε τα κλειδιά του υπουργείου οικονομικών παρέδωσε τα κλειδιά της ελληνικής βουλής και από εδώ και πέρα πια θα αποφασίζουν οι δανειστές νομοθετώντας και τυπικά με προεδρικά διατάγματα τι πρέπει να γίνει στην ελλάδα. από εδώ και πέρα για τα πλεόνασμα για τους φόρους που θα μπαίνουν στα λαϊκά στρώματα για τους φόρους που θα απαλλάσσονται οι πολυεθνικές εταιρείες θα αποφασίζουν οι δανειστές. κύριε Μοσχοβησί, η ευρωζώνη της λιτότητας της ανεργίας των ανισοτήτων και τα μνημόνια τα προγράμματα προσαρμογής που λέτε έχουν κάνει με ευθύνη βεβαίω των ελληνικών κυβερνήσεων που υπογράφουν και εφαρμόζουν μνημόνια το ελληνικό κοινοβούλιο να έχει μόνο διακοσμητικό ρόλο. την απάντηση κύριε μoscovici θα την πάρετε από τον ελληνικό λαό αλλά και από τον γαλλικό λαό και νεολαία που έχει βγει στους δρόμους και στις πλατείες στις ευρωπαϊκές πόλεις. σας ευχαριστώ κυρία πρόεδρε. Κύριε Χοντή, υπάρχει μια μπλε κάρτα από τον κύριο Ζάνη. Την δέχεστε. Παρακαλώ κύριε Ζάνη. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και εσάς που δέχεστε την ερώτηση. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα της αλήθειας επιτέλους και σας ερωτώ ποια θα ήταν η λύση πιστεύετε. Έχουμε ακούσει πολλά για το ποια δεν είναι λέει η λύση, αλλά τι πιστεύετε εσείς ποια είναι η λύση. Και εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω τον κύριο συνάδελφο για την ερώτηση που με έκανε. Κύριε συνάδελφε, η λύση την ξέρουμε. Την ξέρει και η Κομισιόν, την ξέρει και το Eurogroup, την ξέρουν όλοι. Το πρόβλημα του ελληνικού χρέους είναι ένας πολιτικός μοχλός για να επιβληθούν πολιτικές λιτότητε. όταν η ελλάδα βρέθηκε σε πρόβλημα δανεισμού μπορούσαν να επιστρατευτούν οι συνθήκες και όχι να φτιαχτούν οι μηχανισμοί τρόικα ή και να τροποποιηθεί η συνθήκη 136 αν δεν το έχετε παρακολουθήσει για να επιβάλλονται και νομίμως μνημόνια που ζητούν αντιλαϊκά μέτρα. επομένως υπήρχαν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν το θέλησαν και τώρα όπως αποδείχθηκε από τα στοιχεία που έδωσε ο συνάδελφος στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από γερμανικό ινστιτούτο όλο αυτό το δάνειο που πήρε η ελλάδα αυτά τα χρόνια των 220 δισεκατομμυρίων το 210 δισεκατομμύρια πήγε στις γερμανικές και στις γαλλικές τράπεζες και επειδή είμαι παλαιός ευρωβουλευτή κύριε συνάδελφε αυτή ήταν και η ομολογία του προκαθήμενου σήμερα κυρίου μοσχοβησή κυρίου όλι ρεν που ομολόγησε ότι όλα αυτά τα προγράμματα υποτίθεται βοήθεια τη Ελλάδα το κάνουν για να σωθεί η Ευρωπαϊκή, η Ευρωζώνη και οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μου δώσατε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε. Δεν ξεπεράσετε κατά πολύ το χρόνο κύριε Χουντή. Στη συνέχεια ο κύριος Ουτάσον ένα λεπτό παρακαλώ. Δεν μπορώ να αποφύγω να χαμογελάσω όταν ακούω τέτοιες επεξηγήσεις για την ε, ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι είναι πολύ τολμηρές κάποιες τέτοιες τοποθετήσεις. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό βρίσκεται μπροστά σε ένα απίστευτο δίλημα. Έχει τις ε, υποχρεώσεις έναντι των ε, πιστωτών της που δεν δίνουν τις ευκολίες αναδιάρθρωσης του χρέους και έχουμε και τις δεσμεύσει. Ε, Χθε δόθηκε ένα μικρό βήμα ε, που έγινε, αλλά δεν επαρκεί. Κύριε Επίτροπε, δύο πράγματα πρέπει να ζητήσουμε. Να είναι πιο φιλόδοξη η αναδιάρθρωση του χρέου. Από το 2010 γνωρίζουμε ότι δεν είναι βιώσιμο το, το χρέος. Πρέπει το δυνατόν γοργότερα να γίνει η αναδιάρθρωση. Δεύτερον, μια χώρα που έχει ένα επιπλέον ποσοστό πάνω από αυτό το οποίο προβλεπόταν από το πρόγραμμα και το οποίο κράτος βρίσκεται έτοιμο να ε, διαφύγει από την ύφεση πρέπει να βοηθηθεί. Τα αναγκαία ε, συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να πηγαίνουν πιο πέρα από εκείνο που προβλέπεται για να μην είναι εκτός τόπου. Πρέπει να αφήσουμε να αναπνεύσει η ευρωπαϊκή οικονομία και να μην τη στραγγαλίσουμε επιβάλλοντας επιπλέον μέτρα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα από εσά, από τον κύριο Μαζουλίκα. Τη δέχεστε. Παρακαλώ συνάδελφε να θέσετε την ερώτησή uh, Ευχαριστώ, πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφο αναφέρθηκε στην σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνού Νομισματικού Ταμείου, γνωρίζετε ότι η Ελλάδα έχει ε, σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τα δημοσιονομικά τη. Αλλά το ερώτημά μου είναι το εξή. δεν πιστεύετε ότι θα πρέπει να καταλήξει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κοινή πολιτική συμφωνία για το ποια είναι η λύση. Μα αυτή θα ήταν ιδανική κατάσταση αγαπητέ συνάδελφε, αλλά τότε θα έπρεπε να μπορούσαμε να λειτουργούμε και λογικά, δηλαδή αναδιάρθρωση του χρέους Αφενό, πράγμα το οποίο δεν το θέλουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, και από την άλλη όχι άλλα μέτρα λιτότητας, ύφεσιακά μέτρα. Αν ίσιαν αυτά θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε μια ιδανική συμφωνία. Θεωρώ ότι αυτά είναι δύο σημαντικές προϋποθέσεις, αλλά δυστυχώς και οι δανειστέ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θέλουν αυτέ τι δύο προποθέσει. Ο κύριο Τζάνι για ένα λεπτό έχει το λόγο. Χθε ακούσαμε την οδή στη χαρά γιορτάζοντας την 9η Μαρτίου. Νομίζω ότι θα έπρεπε όμως να παίζουμε περισσότερο μια πιο λυπητερή μουσική. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι όλα τα προγράμματα διάσωσης, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, έχουν απετύχει και είχαμε και τη μελέτη Μπάκ, όπου 9,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 216 δισεκατομμύρια των δύο πρώτων πακέτων πήγανε στον ελληνικό λαό. Όλα τα υπόλοιπα χρήματα πήγανε σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και το τρίτο πρόγραμμα επιμένει στα ίδια λάθη. Πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% ενώ δεν προβλέπει καμία ονομασματική απομείωση του χρέους. Πραγματική οικονομική αλλά και κοινωνική τρέλα. Έγκλημα κατά των ίδιων των Ελλήνων είναι αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή ιδιωτικοποίησει άγριε, επιθετικέ, κατάργηση και καταπάτηση πάρα πολλών κοινωνικών δικαιωμάτων, μία ακόμα αναδιάρθρωση του συνταξιδοτικού συστήματος. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το Eurogroup θέλει επιπλέον ένα σύστημα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που δεν καταφέρει η Ελλάδα να πετύχει τους αρχικούς στόχους. Για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι βρίσκεται στη μέγενη η Ελλάδα και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό η χώρα αυτή να απελευθερωθεί από τη μάστιγα του ευρώ. Ο κύριος Βιλίμσκι έχει το λόγο για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ε, αυτά τα οποία λέγονται σήμερα ότι θα λειτουργήσει το πακέτο σταθεροποίησης για την Ελλάδα, ότι θα υπάρξει το τέλος της κρίσης για την Ελλάδα. Αλλά βλέπουμε ότι δεν θα λένε ακόμα τα 28 κράτη-μέλη ότι κάτι θα γίνει, θα υπάρξει μια λύση στην Ελλάδα, θα πάνε χαμένα αυτά τα λεπτά. Βλέπουμε τώρα ότι με κάθε πακέτο η κατάσταση γίνεται χειρότερη και χειρότερη. Το βουνό των χρεών της Ελλάδος διονγκούται συνέχεια, έχει ξεπεράσει το 180% του ΑΕΠ και οποιοδήποτε οικονομολόγο θα σα πει ότι αυτό δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτείται αυτό το, το χρέος. Αυτή τη βδομάδα το Spiegel δημοσίευε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διαχείρισης και Τεχνολογίας λέει ότι 95% των μέσων των κονδυλίων που δόθηκαν στην Ελλάδα τελικά δεν κατέληξαν στην Ελλάδα, αλλά ξαναγύρισαν σε πιστωτές. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα να εξηγιανθεί η Ελλάδα. Και έχουν ουσιαστικά χαθεί όλα αυτά αυτοί οι οποίοι πήραν φτηνά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχουν κερδίσει και δεν έχουν καμία ευθύνη για το κακό το οποίο έχουν προκαλέσει. Το μόνο μάθημα το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή τη διαδικασία είναι να φύγει η Ελλάδα από τη ζώνη του ευρώ για να μπορέσει το μέλλον να γίνει ανταγωνιστική και να εξηγιαστεί. Δεν μπορεί με αυτού του είδους πολιτικές βοήθειες η Ελλάδα να διασωθεί πρέπει να της δώσουμε τη δυνατότητα να έχει και πάλι ένα μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φουντούλης για ένα λεπτό. Για άλλη μια φορά είμαστε θεατές στο ίδιο θέατρο του παραλόγου. Είναι απίστευτε οι καταστάσει που βιώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τέτοια πολιτική αναλγησία και αθλειότητα δεν έχουμε ζήσει ποτέ μέχρι σήμερα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτε, δεμένοι πίσω από το άρμα τη Γερμανία και με επιθύνιο όργανο του στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, γκρέμισαν και τα τελευταία οχυρά τη Ελλάδα καταπάτησαν όλες τις υποσχέσεις τους προς τον λαό προδίδοντας την πατρίδα τους και καταστρέφοντας τον τόπο παραδίδοντάς τον μαζί με τις επερχόμενες γενιές στους γενοκτόνους δανειστές του δουνουτού και κυρίως στους συμμάχους και εταίρους φίλους μας φτωχοποιώντας τον λαό διαλύοντας όλες τις κοινωνικές τάξεις το εμπόριο τη δημόσια υγεία και ό,τι άλλο αφορά τη λειτουργία και την ύπαρξη ενός κράτους τα μνημονιακά δάνεια δεν έσωσαν την ελλάδα αλλά τις ευρωπαϊκές τράπεζες μεταφέροντας τις ζημιές τους στα κράτη μέλη και αυτά με τη σειρά τους έλληνες φορολογούμενους. στον ελληνικό προϋπολογισμό κατέληξαν λιγότερο από το 5% των δανείων ύψους 220 δις ευρώ που δόθηκαν για τη σωτηρία της ελλάδας στα πέντε πρώτα χρόνια των μνημονίων ενώ τα υπόλοιπα πήγαν για τη διάσωση των ευρωπαϊκών τραπεζών σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στη γερμανική οικονομική εφημερίδα handelsblatt σε όλες τις χώρες που επιβάλλατε τη μνημονιακή δίθεν σωτηρία το χρέος τους ως ποσοστό του αεπ το λιγότερο διπλασιάστηκε. στην πραγματικότητα η επιτροπή δεν κάνει δηλώσεις για την πορεία των διαπραγματεύσεων του ελληνικού προγράμματος στήριξης απλά συντάσσει το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Βρισκόμαστε φαίνεται τώρα στον καλό δρόμο, αλλά χρειάζεται να αναμείνουμε πολύ για να μπορέσουν αυτέ οι μεταρρυθμίσει να εγκριθούν στην Ελλάδα από την κυβέρνηση Τσίπρα και είναι κρίμα που χάσαμε τόσο πολύ χρόνο, γιατί θυμόμαστε ότι την εποχή του Αντώνη Σαμαρά είχαμε τόσο μεγάλη πρόοδο στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά θα πρέπει σήμερα να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για τις συγκεκριμένες προόδους οι οποίες έχουν επέλθει και να πούμε ότι ο κύριος αρχιτέκτονας αυτής της πρόοδου είναι ο ελληνικός λαός. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το θάρρος που έδειξαν οι πολίτες της διότι έχουν κάνει μεγάλες προσπάθειες και θυσίες χωρίς να έχουν ένα άμεσο όφελος ε, διέρχονται ακόμα μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Αυτοί καταρχήν χρειάστηκε να υπομισθούν τις συνέπειες της πολιτικής που ακολούθησε η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση της χώρας του σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης. Υπάρχουν ακόμα πολλοί προνομιούχοι και πολλοί που ζουν στην αθλειότητα στην Ελλάδα. Το Eurogroup δεν έδωσε βέβαια την ε, απόλυτη βεβαίως υγεία στην Ελλάδα είναι σαφές ότι η εξυγίανση εξαρτάται από την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Χαίρομαι που το Eurogroup έχει αρχίσει να συζητά και για την δυνητική ελάφρυνση του χρέους. Δεν μπορεί μια χώρα να έχει τόσο υψηλό ποσοστό χρέους και αυτό είναι ακατανόητο και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Μονάχα με σημαντικές όμως μεταρρυθμίσεις θα μπορέσει να γίνει αποδεκτή η απομείωση αυτού του χρέους. Χωρίς την ευρωπαϊκή λοιπόν αλληλεγγύη ακόμα και αν αυτή είναι αντικείμενο κριτικών από πολλούς η η Ελλάδα θα ήταν σε ακόμα πιο σοβαρή κρίση. Κύριε Γκροστέτ, υπάρχει μια μπλε κάρτη από τον κύριο Επιτίδιο. Την δέχεστε? Ο κύριος Επιτίδιος. Ε, ευχαριστώ κύριε συνάδελφε που δέχεστε την ε, παρέμβασή μου. Ε, αναφερθήκατε προηγουμένως σε πρόοδο που είχε σημειώσει η Ελλάδα με διακυβέρνηση της χώρας από τον κύριο Σαμαρά γνωρίζετε ότι και αυτός είναι υπεύθυνο για τη θλιβερή κατάσταση την οικονομική στην οποία βρίσκεται η χώρα μας. Υπέγραψε και αυτός ένα μνημόνιο που υπήρξε προάγγελος του τωρινού μνημονίου. Και πέραν αυτών υπήρξε και ο άνθρωπος ο οποίος καταπάτησε κατά τρόπο απαράδεκτο τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα δημοκρατικά ήθη και έθιμα στέλνοντας παρανόμως στη φυλακή τον αρχηγό και βουλευτές του τρίτου σε πολιτική δύναμη κόμματος. Αυτός είναι ο κ. Σαμάρας τον οποίο εσείς Θαυμάζεται και του οποίου τις ενέργειες επικροτείτε. Ευχαριστώ. Η μόνη διαπίστωση που μπορώ να κάνω είναι ότι την εποχή του κυρίου Σαμαρά παρατηρούσαμε ήδη ανάπτυξη να ξαναρχίσει στην Ελλάδα. Θυμάμαι ότι το είχα αναφέρει και εγώ ίδια Δυστυχώς στη Γαλλία αυτή την ανάπτυξη δεν την είχαμε, ούτε καν αυτή την ανάπτυξη. Είχαν ξεκινήσει μεταρρυθμίσεις. Προφανώς υπάρχουν ε, ευθύνες ε, σε όλους, αλλά το ξεκίνημα της ανάπτυξης ήταν θετικό και κρίμα που χάσαμε χρόνο έκτοτε. Μπούλμαν, λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν δούμε τις αποφάσεις του Eurogroup. Αρχίζω να πιστεύω ότι σιγά σιγά αρχίζει να επανέρχεται η λογική στις διαπραγματεύσεις των Υπουργών Οικονομικών. Ο Επίτροπος ο κ. Μοσκοβίτση θα πρέπει να ξέρει ότι θέλω να τον ευχαριστήσω αυτόν προσωπικά και τους συνεργάτες του για την συνεισφορά που είχε στην επίτευξη αυτής της λογικής. Χρειάζεται τώρα όμως να προχωρήσουμε και να έχουμε αποτελέσματα στις 24 Μαΐου, να έχουμε επενδύσεις, να έχουμε μείωση της ανεργίας, να έχουμε μια πραγματική τομή, να ξεπεραστεί αυτό το οποίο έχει γίνει με την οικονομική κρίση του 2009. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, χρειαζόμαστε απασχόληση για τους Έλληνες. Αγαπητοί συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, άκουσα τρεις εξέχοντες ομιλητές οι οποίοι είπαν ότι η κυβέρνηση τη δική του παράταξη στην Νότια Ευρώπη, οι κυβερνήσει παράταξη στην Νότια Ευρώπη τα έχουν κάνει όλα σωστά και όλε οι άλλε τα έχουν κάνει τελείω λάθο. Αν θέλετε όμω να δείτε ποιο είναι ο κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που επέφερε ο κύριο Σαμαρά, πληροφορηθείτε πρώτα και μετά ελάτε να δείτε αν ευσταθεί το επιχείρημά σα ή αν καταραίει από μόνο του. Εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια οικονομική προοπτική όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για όλη την Νότια Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε έναν τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τι δεξιότητε και τα ταλέντα των ανθρώπων στην Νότια Ευρώπη. Πώ μπορεί να υπάρξει μια κατανομή εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να εκμεταλλεύεται και τι δικέ του δυνατότητε. Ελπίζω θα περάσουμε κάποια στιγμή σε αυτή τη συζήτηση και όχι να μιλάμε μονάχα για το χρέο και την αντιμετώπιση του χρέου. Ο κύριο Σταρμπάτη για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος ε, Πιτέλα είπε προηγουμένως ότι είναι σαν να ξαναβλέπει μια παλιά ταινία να παίζεται πάλι και πάλι. Εμείς ακούμε τα ίδια πράγματα να λέγονται πράγματι και αυτή είναι η ίδια εντύπωση που έχω και εγώ. Και το έχω τονίσει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο ότι ακούω πάντα να υπάρχουν αυτές οι προτροπές και οι επιταγές για το τι θα πρέπει να κάνει κανεί, Ακούω τον κύριο Μοσκοβίτσι να λέει θα κάνουμε αυτό και μετά θα έρθουν οι επένδυσει. μετά θα έρθει η ανταγωνιστικότητα, μετά θα έρθει η ανάκαψη. Τα έχει πει πολλές φορές, τίποτα δεν βγήκε από όλα αυτά. Ο Economist έγραψε ότι η ελληνική οικονομία είναι με απέλπιδα τρόπο μη ανταγωνιστική. Και πραγματικά, ας καταλάβουμε γιατί έχουν μειωθεί οι άνεργοι στη Γερμανία από τα 10% στα 5%. Γιατί όμως το νότο της Ευρώπης από 10% έχουν πάει στα 15% στα 20% οι άνεργοι. Ακριβώς γιατί υπάρχει μια αναντιστοιχία στα επίπεδα τιμών. Αλλά αυτό το κοινοβούλιο δεν αντιμετωπίζει πραγματικά το πρόβλημα αυτό, ότι το ευρώ έχει δημιουργήσει το πρόβλημα αυτό. Ο κύριος Τόρβαλτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τα πράγματα κάπως ευρύτερα. Αν κάνουμε μια ιστορική ανατροπή, θα, ε, αναδρομή, θα διαπιστώσουμε ότι στη δεκαετία του 50 και του 60 η γενική τάση στην Ευρώπη ήταν όλοι να ε, προχωρούν με ρυθμούς 5-6% και βεβαίως αυτό άλλαξε στα μέσα της δεκαετίας του 70. Και βεβαίως αυτό άλλαξε περισσότερο μετά τη διεύρυνση στη δεκαετία του 90. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα πολιτική συνοχή και γι' αυτό χρειάζεται προπολογισμό κατάλληλο για να αντιμετωπιστούν αυτέ οι προκλήσει. Δεν έχει νόημα να μιλάμε στην αίθουσα αυτή για το ποιο έκανε πιο λάθος. Δεν υπάρχει ούτε ένας πολιτικός εδώ ή σε οποιοδήποτε άλλο κοινοβούλιο που να μπορεί να ισχυριστεί ότι έκανε μόνο σωστά πάντα κάποιος κάθε πολιτικός έχει κάτι σε βάρος του. Πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε τις αλληλοκατηγορίες και να πρέπει να ε, προχωρήσουμε με ένα νέο προπολογισμό για να διορθωθούν τα προβλήματα των χωρών της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν πραγματικά επικίνδυνες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Σακοράφα για... Χαίρομαι που οι περισσότεροι αναγνωρίζετε σήμερα εδώ ότι πραγματικά έχει διαπραχθεί ένα έγκλημα εναντίον του ελληνικού λαού αλλά κύριοι συνάδελφοι και οι χθεσινέ πολιτικέ εξελίξεις φανερώνουν για μια ακόμα φορά ότι στην ευρώπη σήμερα υπάρχει μια κυρίαρχη δύναμη που αδιαφορεί για τη δημοκρατία για τα δικαιώματα και τι ανθρώπινε ζωέ. επιβάλλει κόφτε, μνημόνια και οδύνη. υπάρχει επίση στην ελλάδα ένα πρόθυμο Πρωθυπουργό που εφαρμόζει αυτή την πολιτική δηλώνοντα ότι ο ριζοσπαστικό εναλλακτικό δρόμο είναι αυταπάτη. υπάρχει όμω στην ευρώπη και μια δύναμη καταγεγραμμένη και εδώ μέσα που δεν έχει αυταπάτες για τα μνημόνια και υπερασπίζεται το δρόμο τη δημοκρατία και τη κοινωνική δικαιοσύνη. Υπάρχει στην Ευρώπη και ένα λαό που χωρί αυταπάτες δεν υπέκυψε στου εκβιασμού του Ευρωπαϊκού Διευθυντηρίου και είπε όχι στη διάσωση των τραπεζών επιλέγοντα τη δική του διάσωση. Υπάρχουν λοιπόν και δύο ειδών αξιολογήσει αυτή που μετράει την υποταγή και την κατάρρευση τη ελληνική κοινωνία σαν κέρδο των τραπεζών και αυτή που μετράει την αντίσταση του ελληνικού λαού σαν κέρδο τη Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή τη συγκρουσιακή ευρωπαϊκή πραγματικότητα, καθένας μας αξιολογείται από το ποιον υπερασπίζεται και για ποια Ευρώπη παλεύει. Thank you. Madame one minute. La présidente, Monsieur le Commissaire, Πρόεδρε, η εφημερίδα Handelsblatt πριν λίγο ανέφερε ότι το 95% του χρέους της Ελλάδος πήγε στις ευρωπαϊκές τράπεζες, στους πιστωτές της. Η Ελλάδα πληρώνει πολύ ακριβά την πρόσβαση στο υπόλοιπο 5%. Τα μέτρα λιτότητας που πέρασε η κυβέρνηση Τσίπρα θα έπρεπε να έχουν ως αντιστάθμισμα την επανεξέταση του ελληνικού χρέους. Χθε ε, το Eurogroup δειλά ξεκίνησε τη σχετική συζήτηση καθυστερώντας υπάρχει το ενδεχόμενο να παραπεμφθούν η συζήτηση του χρέου στο τέλος του προγράμματος. Πώς μπορεί να προβλέψει το μέλλον και να επενδύσει στο μέλλον μια οικονομία υπό τις συνθήκες αυτές. Η απουσία διεξόδου δημιουργεί κοινωνική αγωνία. Το 2018 όταν η ελληνική οικονομία έχει υποστεί τις επιπτώσεις του νέου προγράμματος λιτότητας, η παλιά εποχή θα είναι, θα είναι μόνο μία μνήμη. Θα επιμείνουμε στο λάθος, θα πρέπει ο ελληνικός λαός να δεν θα υπάρχει ούτε κέρδος για τον ελληνικό λαό, ούτε, για, ούτε αποζημίωση για τους πιστωτές της Ελλάδος. Γιατί επιμένετε στον δρόμο αυτό, κύριε Επίτροπε. Κύριε Φων Στόρκ. Δεν είναι παρούσα όμως. Ο κύριος Φιλιππό. Για 1,5 λεπτό. Την προηγούμενη Τετάρτη το Handelsblatt, η γερμανική αυτή οικονομική εφημερίδα, που έχει σοβαρούς οικονομολόγους, είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είπε ότι η βοήθεια προς την Ελλάδα δεν πήγε στον ελληνικό λαό, αλλά πήγε στις τράπεζες. Λιγότερο από 5% από τα συνολικά ποσά που δώσαμε όλοι μας πήγανε στην ελληνική οικονομία. Το τίμημα αυτού του 5% ήταν για τους Έλληνες μια απόλυτη άρνηση δημοκρατίας και μια μεγάλη βία προς αυτούς. Από το 2010, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεπε την χρεοκοπία της Ελλάδος, εσείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργήσατε μια πυραμίδα πόντσι για να σώσετε τις τράπεζες και όχι το λαό, για να μπορέσει να ε, ξαναπληρώσει το χρέος του, ο ελληνικός λαός έπρεπε να δανείζεται όλο και περισσότερο. Αποφασίσατε να τιμωρήσετε με μια τρομερή βία και ομότητα τον ελληνικό λαό όταν προσπάθησαν να επιλέξουν μια άλλη δημοκρατική οδό εκλέγοντας τον κύριο Τσίπρα ή στη συνέχεια λέγοντας όχι στο δημοψήφισμα για το σχέδιο διάσωση. Υποβάλλατε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος δεν είχε το θάρρος να αντισταθεί και δεν είχε το θάρρος να ακολουθήσει την έξοδο από το ευρώ σε μια τέτοια διαδικασία βασανισμού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί τον εκβιασμό τους για την παροχή ρευστότητα. Έχετε επιβάλει μια τέτοια κατάσταση στο λαό των Ελλήνων, ενώ είναι οι δικές σας επιλογές που φταίνε για όλα αυτά. Οι λεγόμενοι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να σηκωθούν από τους τάφους τους και να δουν ποια θα έπρεπε να είναι η πραγματική Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κύριος Μούρεσαν, για ένα λεπτό και μισό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι Επίτροπε. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα είναι αποτέλεσμα πολιτικών δράσεων που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση από τότε που ξεκίνησε. Η Ελλάδα έβγαινε από την κρίση το δεύτερο εξάμεινο του 2014 με οικονομική ανάπτυξη άνω του 2% για το 2015 και πλεόνασμα. Όλα αυτά τέθηκαν σε κίνδυνο από την παρούσα κυβέρνηση πέρυσι που έκλεισε τις τράπεζες για τρεις εβδομάδες χωρίς οικονομία. Ποιο είναι ο δρόμο προ τα εμπρό τώρα, κατά την άποψή μου, είναι οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι μεταρρυθμίσεις. Μία λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση προ όφελο των πολιτών μια μεγαλύτερη και πιο ευέλικτη αγορά εργασίας που θα επιτρέψει στους νέους να βρουν δουλειά και που θα διευκολύνει και να διευκολύνεται η ανάληψη ε, από τους νέους ε, νέων επιχειρήσεων. Καλύτερη παιδεία, σωστό επιχειρηματικό πλαίσιο. Αυτό θα οδηγήσει σε επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Τα μέτρα αυτά δουλεύουν. Τα είδαμε στην Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ισπανία. Το μόνο σημείο όπου απέτυχαν ήταν στην Ελλάδα. Αν η οικονομία ωστόσο δεν είναι ανταγωνιστική, τα υπόλοιπα ε, ε, θα διορθωθούν. Δεν θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη, με άλλο τρόπο δεν θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των επενδυτών και δεν θα μεταρρυθμιστεί η οικονομία. Ευχαριστώ. Η Μπερές. 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, για να δώσουμε μια ποικιλία σε αυτά που λέμε για την ε, ε, κατάσταση Ελλάδος, μπορούμε να καταλήξουμε στα εξή συμπεράσματα από τη χθεσινή συνάντηση του Eurogroup. Το ένα είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση ε, έχει κάνει σοβαρή προσπάθεια μεταρρυθμίσεων και αυτό πρέπει να το χαιρετήσουμε. Την Κυριακή ψηφίστηκε ο νόμος για την μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος με συμπέρασμα 3 ε, δισεκατομμύρια το χρόνο ε, οικονομίες. Ο Πρωθυπουργός κύριος Τσίπρας έκανε αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Δεύτερον, το θέμα του ελληνικού χρέους ε, έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται αλλά πρέπει και εμείς να τηρήσουμε την πρότασή μας ε, του 2012. Και το τρίτο είναι ότι πρέπει να πάρουμε μαθήματα από, τον, ε, από την αισιοδοξία με που οφείλεται σε εξαιρετικές, εξαιρετικά ξεκάθαρες πράξεις και στις 24 Μαΐου θα πρέπει να δοθεί ε, μια διαβεβαιότητα έτσι ώστε οι επενδύσεις να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα γιατί τις έχει μεγάλη ανάγκη και αυτό θα βοηθήσει και την Ελλάδα αλλά ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ε, Ένα λεπτό, ο κύριος Μονό παρά την λαμπρή συμφωνία του 2015, του Αυγούστου 2015, τίποτα δεν λύθηκε στην Ευρώπη. Όπως καταγγέλει το Εθνικό Μέτωπο, η ευρωλιτότητα δεν δίνει αποτελέσματα. Καθιστά αδύναμη, αδύναμο το, την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Η Ελλάδα είναι ένα σύμπτωμα του καρκίνου του ενίου νομίσματος. Για ένα πατριώτη το χρέος είναι χρέος. Μία, ε, ένα haircut θα είναι ανεύθυνο γιατί θα είναι μερική χρεοκοπία που θα ανατινάξει όλη την, ε, την ισορροπία του ευρώ. Αντίθετα, οι υπεύθυνοι πιστωτές πρέπει να μπορέσουν να επιτρέψουν στην Ελλάδα μια νέα αρχή, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχουν τρεις βασικοί όροι. Πρώτον, κυριαρχία νομισματική, βγαίνοντας από το ευρώ, ούτως ώστε να αποπληρώσει τμήμα του χρέους της. Δεύτερον, την επιστροφή των αποζημιώσεων από τη Γερμανία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και αποφυγή μιας οικονομικής κρίσης και μιας οικονομικής κρίσης σώζοντας και τη δημοκρατία. Ο κύριος Κίρτσος, 1,5 λεπτό στην ελλάδα έχουμε καλά αλλά έχουμε και δυσάρεστα οικονομικά νέα. τα καλά νέα είναι ότι η κυβέρνηση τσίπρα έχει εγκαταλείψει τη στρατηγική της αντιπαράθεσης με την ευρωζώνη και κάνει την αναγκαία προσπάθεια προσαρμογής. άρα δεν θα έχουμε επανάληψη της κρίσης του. 2015. δυστυχώς όμως υπάρχουν και δυσάρεστα νέα. πρώτον είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε ακριβά το λογαριασμό του αποτυχημένου ριζοσπαστικού πειράματος τσίπρα βαρουφάκη του 2015 δεύτερον το μείγμα οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση σύριζα δίνει την έμφαση στην εξοντοτική φορολόγηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και των νοικοκυριών με αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέα προβλήματα στη λειτουργία της οικονομίας. τρίτον ύστερα από απέτηση του διεθνούς νομισματικού ταμείου η κυβέρνηση τσίπρα δέχθηκε τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρέμβασης και την προετοιμασία των λεγόμενων προληπτικών μέτρων για το. 2018 έτσι στέλνει το μήνυμα ότι το ελληνικό πρόγραμμα δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστο και καταργεί τον εμπροστοβαρή χαρακτήρα του τρίτου προγράμματος και του σχετικού μνημονίου με αυτόν τον τρόπο τα κάνει λιγότερο αποτελεσματικά και λιγότερο αναπτυξιακά. τα παραπάνω αποδεικνύουν το τεράστιο κόστος του αριστερού λαϊκισμού. ο σύριζα προκάλεσε πρόορε εκλογές στα τέλη του 2014 εμποδίζοντα την έξοδο τη Ελλάδα από το μνημόνιο με την εφαρμογή των τελευταίων μέτρων ύψους 1,2 δις ευρώ. όμως η κυβέρνηση τσίπρα έχει ήδη εφαρμόσει ανακοινώσει ή προγραμματίσει μέτρα δεκαπλάσιου ύψους. αυτό τα λέει όλα για τον αριστερό λαϊκισμό. ελπίζουμε το πάθημα του ελληνικού λαού να έχει γίνει μάθημα και για τους ευρωπαϊκούς λαούς. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ενώ κορυφώνεται το δράμα των Ελλήνων με νέα απελπιστικά μέτρα λιτότητα, νέε περικοπέ συντάξεων και την πιο άγρια φοροεπιδρομή στου πιο φτωχού από την πιο ανάλγητη εθνικολαϊκιστική κυβέρνηση τη μεταπολίτευση, ορισμένοι πανηγυρίζουν τη βολική και εξυπηρετική αυτή πολιτική ως λευκή επιταγή στην τρόικα και σε κάθε απέτησή τη. μερικές φορές η υποκρισία περισσεύει και ανάμεσά μα μόνο που σήμερα το άλοθη για τον δράκο του δούνου του μας τελείωσε καθώς από την ευρωπαϊκή ένωση έγινε αποδεκτή μια συμφωνία που εκδικείται τους πιο αδύναμους πολίτες χωρίς πραγματικές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις. η πολιτική σόιμπλε είναι αυτή που εξυπηρετείται απολύτως και μεταθέτει την όποια ελάφρυνση των στόχων για το 2018 και βλέπουμε και ενώ κάποιοι όψιμοι φίλοι εθελοτυφλούν και στο απόλυτο ξεπούλημα των περιουσιών των ελλήνων σε ξένα φαντ και κερδοσκόπου από τη συγκυβέρνηση σύριζα ανέλ τη σημαία της ε, αλληλεγγύης ας την αφήσουμε για όταν πραγματικά αποφασίσουμε να ενδιαφερθούμε για τους πολίτες και όχι για του αριθμού και τις σημαίες αριστεροσύνης. ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο Eurogroup ο κύριος ε, Σόιμπλε είπε ότι η Ελλάδα έπρεπε να πάρει μια σκληρή απόφαση. Ο στόχος είναι να προχωρήσει. Η Ελλάδα έκανε τις αναγκαίες δημοσιονομικές τροποποιήσεις, ωστόσο ο στόχος πέρσι ε, άλλαξε. Μετά από τις κακές αποφάσεις της Ελλάδος του παρελθόντος μπορούμε να μιλούμε ίσως και για ε, ελάχιστα ρεαλιστικές απαιτήσεις των χωρών της Ένωσης. Η Κριστίν Λαγκάρντ είπε η ίδια ότι το 3,5% πλεόνασμα δεν είναι ρεαλιστικό. Το Δέλτα Νι Ταφ αναγνώρισε ότι ήδη το 2010 πρέπει να μιλήσουμε για ελάφρυνση του χρέους. Είναι καιρός να κάνουν μια αυτοκριτική και οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κυρώσεις για τις οποίες μίλησε ο Σόιμπλε δεν ισχύουν πλέον. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να διδαχθούμε από τα λάθη μας και πρέπει να βοηθήσουμε την Ελλάδα να αποκατασταθεί. Ο κύριος Κύρικος, ένα λεπτό. Το χθεσινό Eurogroup μας απέδειξε πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και οι ελληνικές κυβερνήσεις συνεργάζονται αδιατάρακτα. Έξι χρόνια κρίση, τρία μνημόνια, δώδεκα θετικέ αξιολογήσει και πάντα έρχεται μια κυβέρνηση η οποία θριαμβολογώντα μα λέει πω οι αριθμοί θα ευημερήσουν αύριο και το μόνο που βλέπουν οι πολίτε είναι καινούργια άμεση και έμεση φόρη. Γιατί άργια συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί οι μεν ευρωπαϊκοί θεσμοί, ξεχνώντα την ανάπτυξη, σχεδιάζουν μόνο δημοσιονομικού στόχου που καταραίουν επειδή δεν έχουμε ανάπτυξη. Οι δε κυβερνήσει αρνούνται τι μεταρρυθμίσει ακριβώ γιατί μπορεί να απειλούσαν το βαθύ ελληνικό πελατειακό κράτο. Όμω, 12 θετικέ αξιολογήσει μα έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχει διέξοδο αν δεν γίνουν σημαντικέ μεταρρυθμίσει που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστο, όπω η ανανέωση του δημόσιου τομέα και τη επιδοτούμενη γεωργία, η μείωση φαρμακευτική δαπάνη, η μείωση του χρόνου απονομή δικαιοσύνη, το σταμάτημα του λαθρεμπορίου καυσίμων το σταμάτημα της διαφθοράς στις δημόσιες δαπάνες. Αυτά ακριβώς που πέντε χρόνια δύο κυβερνήσεις δεν άγγιξαν και δεκαπέντε μήνες η τωρινή κυβέρνηση δεν έχει καν ξεκινήσει. Thank you. Mr. Fernandez, one minute. Κύριος Φερνάντες, για ένα λεπτό. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Φερνάντες. Oh, it's working. Perfect. Muchas gracias. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μοσκοβίτση για το έργο του εδώ και πάνω από ένα χρόνο μετά από το γεγονός ότι πέρσι το φθινόπωρο είδαμε να πέρσι το καλοκαίρι μάλλον είδαμε να γίνεται αυτό το δημοψήφισμα όταν ήμασταν σχεδόν έτοιμοι να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Έχουμε χάσει σχεδόν ένα χρόνο και επιτέλους έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία η οποία είναι λογική και εγώ βέβαια όπως και η κυρία Καηλή, όπως οι άλλοι συνάδελφοί μου στη σοσιαλιστική ομάδα το διαμφισβητούμε. Δεν ξέρουμε πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε την κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά έχουμε φτάσει σε μια συμφωνία λογική. Θέλω λοιπόν να τονίσω ότι είναι απαραίτητο να γίνουν οι μεταρρυθμίσει, οι πραγματικέ αυτέ μεταρρυθμίσει που θα δημιουργήσουν δυνατότητα ανάπτυξη στον εξαγωγικό τομέα, να υπάρξουν αυτέ οι μεγάλε μεταρρυθμίσει που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και όπω έλεγε και ο κύριο Τάγκ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ήδη από τώρα το θέμα του χρέου. Έχει γίνει η δέσμευση, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ περισσότερα, γιατί δεν μπορούν οι πολίτε τη Ευρώπης, της Ελλάδος να πλήττονται με ακόμα περισσότερε περικοπέ, γιατί θα χάσουν κάθε ιδέα και κάθε εμπιστοσύνη στην Ευρώπη έτσι. Ο κύριος Μαυρίδη, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Μοσκοβισή, σήμερα έχουν λεχθεί πάρα πολλά για το παρελθόν και λιγότερο για το παρόν και το μέλλον το ερώτημα είναι πολύ απλό έχει συμφωνηθεί ένας οδικός χάρτης που έστω και καθυστερημένα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση της ανάπτυξης. το δεύτερο που έχουμε μπροστά μας είναι ότι παρά τα όποια λάθη έχουν γίνει έχουν γίνει και σοβαρές μεταρρυθμίσεις. το ερώτημα λοιπόν είναι απλό για όλους μας θα βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό ο οποίος υποφέρει και έκανε θυσίες ως μέλος αυτής της οικογένειας; θα βοηθήσουμε τον ελληνικό λαό που ανοίγει τις αγκάλες του στους κατατρεγμένους την ίδια ώρα που πολλά κράτη μέλη στείνουν φράχτες. όσο για το χρέος το απαντώ όσο πιο απλά μπορώ χωρίς ελάφρυση του χρέους στο βαθμό που να μετατραπεί σε βιώσιμο ανάπτυξη μέσω ορθολογιστικών επενδύσεων δεν πρόκειται να προκύψει. επενδύσεις σε μια οικονομία με χρέος εκτός ελέγχου δεν γίνονται. όσο για το διεθνές νομισματικό ταμείο που ζητά λιγότερη λιτότητα αλλά απαιτεί προληπτικά μέτρα λιτότητας αδυνατό να κατανοήσω τη λογική τους. Thank you. And now this concludes the debate with the representatives of political groups. Now we move to the kitchen. Έχουμε κλείσει τη διαδικασία συζήτησης. Περνάμε στην διαδικασία καστία με πρώτη την κυρία Σπυράκη. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε Μοσχοβησή, χθε το Eurogroup επανέλαβε την απόφαση για το χρέο από τον Νοέμβριο του 2012, όμω, με προστιθέμενα και αυξημένα μέτρα με αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομική διόρθωση. είναι μια υπόσχεση που εκκρεμεί τέσσερα χρόνια και στη διαδρομή μόνο από τον ιανουάριο του 2015 έχουν φύγει από τις τσέπες των ελλήνων 9 δισεκατομμύρια ευρώ παράλληλα έχετε κι εσείς ευθύνη ως δανειστές αφού επιτρέπετε ένα μείγμα πολιτικής που βασίζεται σε περισσότερη φορολογία σε περισσότερες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών που ευνοούν και τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος η ελλάδα δεν χρειάζεται άλλα προγράμματα χρειάζεται μια άλλη πολιτική με λιγότερους φόρους με λιγότερες δαπάνες χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση που θα προχωρήσει γρήγορα σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να μην ξανασυζητήσουμε εδώ το ελληνικό πρόβλημα για να είναι η ελλάδα πρωταγωνιστής στην καρδιά της ευρωζώνης και βεβαίως και πρώτα απ' όλα και κυρίως εσείς να τηρήσετε τις υποσχέσεις σας που εκκρεμούν εδώ και μια τετραετία. σας ευχαριστώ ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι επίγον να βγούμε από μια αποκλειστικά λογιστική προσέγγιση δίνοντας μια προοπτική στην Ελλάδα, ακόμη περισσότερο στον ελληνικό λαό. Πρέπει να δράσουμε προς δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Βεβαίω χρειάζονται μεταρρυθμίσει ουσία το ξέρουμε όλοι, στο κράτο, στη διοίκηση, στην δικαιοσύνη, στην υγεία. Προσθέτω ωστόσο ότι αν είχαν γίνει μεταρρυθμίσει πριν, δεν θα έπρεπε να τι κάνει σήμερα ο κ. Τσίπρα. Πρώτο θέμα. Δεύτερον, ναι, πρέπει να αναδιαρθρώσουμε το χρέος, να το επαναπροσανατολίσουμε. Χρειάζεται στην πράξη να θέσουμε την βοήθεια σε επικοδομητικά αναπτυξιακά έργα. Πρέπει η Ελλάδα να ξαναχτίσει τη βιομηχανία της, την γεωργία της, να αποκτήσει νέους ε, δρόμους ε, στις ανανεώσιμες για παράδειγμα. Και τέλος, κλείνοντας, αντί να δακτυλοδεικτούμε την Ελλάδα και τους Έλληνες, θα έπρεπε να δούμε και λίγο τη δική μας πλευρά προσπαθώντας να διαμορφώσουμε ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ανδρουλάκης. Καθώς από το Eurogroup, αλλά βαρύ το τίμημα για την ελληνική οικονομία. Περισσότεροι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές στις παραγωγικές δυνάμεις δεν προϊονίζουν τη μείωση της ανεργίας που είναι το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα της Ελλάδας διαγενειακή αδικία καθώς οι νέοι όσοι τουλάχιστον από αυτούς εργάζονται στην ελλάδα θα πληρώσουν μεγαλύτερες εισφορές για μικρότερες συντάξεις. η ευθύνη βαραίνει του δανειστές και την ελληνική κυβέρνηση. το όλημα στρατηγικής για καλύτερες μέρες αναδεικνύει την απουσία οράματος. αυτό είναι ο κύριος λόγος που όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι αδυνατούν να εντοπίσουν στη σημερινή ευρώπη τις αρχές και τις αξίες που γιορτάσαμε μόλις χθε. τέλος αν πιστεύετε εδώ μέσα κάποιοι πραγματικά ότι το δούνου του είναι εμπόδιο σε μια δίκαιη λύση για το χρέο το ελληνικό αλλά και μια πιο δίκαιη αντιπολιτική λιτότητα για το ελληνικό πρόγραμμα και θέλουμε την αποχώρηση τότε α ψηφίσουμε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να φύγει το δούνου του από το ελληνικό πρόγραμμα εκτό βέβαια αν το χρησιμοποιείτε μόνο ω άλοθη. Επειδή προέρχομαι από την Ιρλανδία, έχω μεγάλη κατανόηση για το δράμα του ελληνικού λαού και έχουν υποφέρει όπως είχαμε υποφέρει και εμείς. Ακούσαμε τα ίδια επιχειρήματα. Μας είπαν ότι δεν μπορούμε παρά να χρεοκοπήσουμε, θα βγούμε εκτός από την Ευρωζώνη αν δεν δώσουμε τα λεφτά στις τράπεζες. Μερικά χρόνια αργότερα, χάρη στην κυβέρνησή μας και χάρη στις θυσίες του Ιρλανδικού λαού, είμαστε όμως τώρα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα στην Ευρώπη και ελπίζω θα μπορέσουμε να το πούμε αυτό και για την Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Την τελευταία φορά που μίλησα εδώ ήμουνα πολύ επικριτικός για τον ε, Πρωθυπουργό της ε, Ευρώπης και του, της Ελλάδος και του έχω ζητήσει να δείξει περισσότερο ευρωπαϊκό πνεύμα και μεγαλύτερη ηγετική δύναμη. Έχει αλλάξει. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορεί κανείς να αποδεχθεί τα ασφάλματά του και να σταματήσει την πολιτική επίδειξη του Υπουργού Οικονομικών του, του κ. Βαρουφάκη στο παρελθόν. Θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να είμαστε εύκαμπτοι και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ελληνική κυβέρνηση ώστε να προχωρήσουμε στην απαραίτητη ανάκαμψη και να τρέψουν και αυτοί τους καρπούς που έχουμε τρέψει εμείς στην Ιρλανδία. Thank you. Mr. Ευχαριστώ κ. πρόεδρε. Ίσως πρέπει να αποδεχθούμε ότι η Ένωση έκανε λάθος επιμένοντας την πολιτική λιτότητας. Ίσως ε, πρέπει να πούμε ότι το αντιστάθμισμα που ζητούσαμε από τις Ένωσες ήταν υπερβολικά και τα μέτρα που είχαν θετηθεί ανεπαρκή για να ε, ξαναπάρει μπρο η ελληνική οικονομία. Ωστόσο, δεν, θέλει, δεν φαίνεται να θέλει να αλλάξει η στρατηγική το Eurogroup. Ήδη ακόμα απαιτεί νέα μέτρα, έναν αυτόματο μηχανισμό αντιστάθμισης που θα κινητοποιηθεί αν υπάρχει, κόβοντας δαπάνες, αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι του προπολογισμού που περιγράφονται στο πρόγραμμα. 3,5% ε, πλεόνασμα κατά βάση στο 2018. Ε, από την άλλη αγνοείται το αίτημα της Ελλάδος για την ε, επιμήκυνση των ε, ε, για την μείωση του χρέους με απλή επιμήκυνσή του. Η Αθήνα έκανε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, φορολογικό νομοσχέδιο. Θα πρέπει να βοηθήσει και το Eurogroup κάνοντας βιώσιμο το ελληνικό χρέος και όχι απλά Κύριε Καπούτο, μπορείτε να, μιλάς, να μιλήσετε λίγο πιο αργά. εκείνο mm. την περίοδο για την οποία η Αθήνα δεν θα, μπορούσε, δεν θα έπρεπε να πληρώνει τόκους. Ευχαριστώ. Σας έχασα. Σας έχασα μεταφραστές κύριε Καπούτε. Ευχαριστώ. Κύριε Κεκόνεν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ελλάδα έχει αυτή την στάση εδώ και πολύ καιρό. Και γι' αυτό το κόμμα μου το 2010 αντιτάχθηκε στο σχέδιο διάσωσης της Ελλάδας. Αυτό ήταν ένα πακέτο για τις γερμανικές και τις γαλλικές τράπεζες βέβαια και όχι για την Ελλάδα. Σε μια δημοκρατία η πλειοψηφία πρέπει να αποφασίζει αυτό το οποίο έγινε το 2010. Εμείς ουσιαστικά ήμασταν η μειοψηφία στο Φιλανδικό Κοινοβούλιο και αναγκαστήκαμε να δεχτούμε την άποψη αυτή που, τις πλειοψηφίας που οδήγησε σε κανόνες που όλοι τους παρέκαμψαν. Έχουν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, αλλά όχι όλες οι απαιτούμενε. Θα πρέπει να δούμε και εμείς την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μερικές φορές δεν μπορούμε να πιστεύουμε όλα αυτά τα οποία μας λέγονται. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει τα απαραίτητα μόνη της προτού να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για να την βοηθήσουμε περισσότερο. Και αν η Ελλάδα φύγει από το ευρώ θα μπορέσει να λύσει όλα τα προβλήματά της και να βελτιώσει την κατάσταση των φτωχότερων πολιτών. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και η πρόεδρος. Ο κ. Χρυσόγονος, τελευταίος ομιλητής. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup έγινε αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους προϋποθέτει τη λήψη μέτρων σε βραχυπρόθεσμο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. όλα αυτά είναι θετικά αρκεί να μετουσιωθούν σε συγκεκριμένες και αποτελεσματικές δράσεις. πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι ούτε η ελλάδα ούτε κανένα άλλο κράτος εκτός ή εντός ευρώπης δεν μπορεί να επιτύχει πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος ετησίως σε βάθος δεκαετιών. η ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν πρόκειται να επανέλθει σε πρωτογενή ελλείμματα αλλά και τα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης πρέπει να βρουν τρόπο για να περιοριστεί το βάρος του ελληνικού χρέους σε τέτοια επίπεδα ώστε να μπορέσει να αναχρηματοδοτηθεί από τις κεφαλαίες αγορές. μια ρεαλιστική και γενναία αναδιάρθρωση θα είναι τελικά προς όφελος τόσο της ελλάδας όσο και των δανειστών της. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελειώνει διαδικασία Catch the Eye και δίνω το λόγο στον κύριο Μοσκοβιτσί για να κλείσει το, τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν το λόγο στη συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι ήταν μια χρήσιμη και καρποφόρα συζήτηση. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο να σας απαντήσω γιατί είναι πολύπλοκες και ποικίλε οι απόψει οι οποίε διατυπώθηκαν. Απλώς θα πρέπει να διαπιστώσω ότι έχουν γίνει λάθη και προφανώς ε, θα πρέπει να βρούμε και τις ε, ευθύνε αυτών που έπραξαν τα σφάλματα αυτά. Μετά από τα 6-7 χρόνια βλέπουμε κάθε μορφή ελλείψεις ε, στην πρόοδο που έχουν γίνει. Έχω, προσπαθώ να δω με κάποια απόσταση όλα αυτά τα ζητήματα, ιδίως στο διάστημα που ήμουν εγώ ο αρμόδιος επίτροπος για τα θέματα αυτά, αλλά και στο παρελθόν όταν ήμουν απλός υπουργό οικονομικών της χώρας μου στο Eurogroup, που εξακολουθεί να είναι η χώρα μου, η Γαλλία λοιπόν. Είναι πάνω από τέσσερα χρόνια λοιπόν που εγώ συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις για την Ελλάδα. Αυτό για το οποίο μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι είναι κατανεμημένες οι ευθύνες, επιμερισμένες οι ευθύνες για τα θέματα αυτά. Έγιναν σφάλματα σε πολλές χρονικές στιγμές από όλες τις ε, ελληνικές κυβερνήσεις στη στιγμή που βρισκόμαστε τώρα βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική καμπή και είναι η κατάλληλη στιγμή να έχουμε μια συνένεση για την ανάγκη διατήρησης της αλληλεγγύης με την Ελλάδα που όλοι αναγνωρίζουν τις προσπάθειές της. Και νομίζω ότι υπάρχει μια λογική σκέψη που θα πρέπει να κάνουμε. Δεν, πρόκειται κάποιος από εμά να πει στην Ελλάδα αν θέλει να μείνει ή όχι στη χώρα του, στην ζώνη του ευρώ. Είναι φανερό ότι ο ελληνικός λαός θέλει να μείνει και αυτή είναι η επιλογή που έκανε. Διατηρεί τη φιλοδοξία να παραμείνει η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ. Αυτό φάνηκε σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Όλα τα μέλη τώρα του Eurogroup είναι άνθρωποι που προέρχονται από όλες σχεδόν τις πολιτικές οικογένειες που είναι εδώ. Είναι άνθρωποι που έχουν διαφορετικές πολιτικές ευαισθησίες. Αυτό το οποίο επιτύχαμε χθε μετά από πάρα πολλή εργασία είναι να ξεπεράσουμε ένα συγκεκριμένο ορόσημο. Το ορόσημο όπου ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων το οποίο είναι εν εξελίξη και είναι <clears throat> στεναρό μπορεί να γίνει αποδεκτό από όλους μας και μπορεί να αποτελέσει τη βάση σε μια επιστροφή της εμπιστοσύνης και της ανάπτυξης στην, Ευρώπη, στην Ελλάδα και να φέρει επενδύσεις για να βοηθήσει αυτόν τον ελληνικό λαό ο οποίος έχει υποστεί τα πάντινα από την κρίση. Και οφείλουμε στον ελληνικό λαό αυτή τη βοήθεια. Δεν μιλάω για κάποια πολιτική παράταξη, δεν μιλάω για τις αρχές της προηγούμενης ιστορίας. Εμείς έχουμε εργαστεί με όλες αυτές τις προηγούμενες κυβερνήσεις για να μπορέσουν να εφαρμοστούν αυτές οι δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή έχει οδηγήσει και σε πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που θα τις λάβει υπόψη και το Eurogroup της 24ης Μαΐου. Έχουμε καταγράψει όλες τις παρατηρήσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί βέβαια ο καθένας να ζητάει, να, να θέλει μάλλον να ακολουθήσει μία κατεύθυνση ή μία άλλη κατεύθυνση, αλλά θέλω να σας πω που είναι η πρώτη φορά που όλα αυτά τα θέματα έρχονται από κοινού και συζητιούνται η συζήτηση για τις διαφορετικές αλλαγές που βρίσκονται μέσα σε μια φιλόδοξη ε, φιλόδοξη δέσμη, επίσης ο μηχανισμός ε, έκτακτης ανάγκης, ο κόφτης ο λεγόμενος, για να μπορέσει να υπάρξει μια λύση σε δύσκολες καταστάσεις και επίσης είναι η πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2004, ακριβώς επειδή υπάρχει ένα στεναρό πακέτο, αρχίσουμε να συζητάμε και για το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού ε, χρέους. Θέλουμε λοιπόν να το πράξουμε αυτό Νομίζω ότι χθε περάσαμε ένα σημαντικό ορόσημο, το επαναλαμβάνω. Ελπίζω ότι στις 24 Μαΐου θα μπορέσουμε να καταλήξουμε και σε μια συμφωνία όσο το δυνατόν ευρύτερη, τουλάχιστον στα δύο βασικά θέματα ή δυνατόν για το σύνολο των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την κατάσταση της Ελλάδας. Άκουσα το ομιλητές από πολλές χώρες που έχουν περάσει και αυτές προγράμματα προσαρμογής και που θα θέλανε και αυτοί να δουν την Ελλάδα να βγαίνει από τα προγράμματα λιτότητος ε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω περάσει ίσως 60, 70, 80 συνεδριάσεις του Eurogroup για τα θέματα αυτά. Ελπίζω κάποια στιγμή σε ένα Eurogroup να μπορέσουμε να πούμε ορίστε η Ελλάδα έχει βγει από το πρόγραμμα προσαρμογής. Θα είναι λοιπόν μια χώρα ακόμα που θα έχει επιτύχει στις μεταρρυθμίσεις της, θα έχει ξαναβρει την ανάπτυξη και αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι η θέληση πιστεύω όλων ανεξάρτητα από πολιτική παράταξη ανεξάρτητα από τις ε, θέσεις που έχουν. Νομίζω ότι είναι το κοινό σας συνέστημα και σας ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ κύριε